Αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να καθίσετε για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας από χθε. Πριν να ξαναρχίσουμε ε, θα ήθελα να σας υποδείξω ότι σε αυτή την Επιτροπή μιλούμε πάντα για τα προσόντα των νέων. Λοιπόν, σας ε, προσκαλώ στη... να πάτε στην έξοδο της αίθουσας όπου υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σας ε, προτείνεται από μια ε, νέα νεαρή φοιτήτρια η οποία φυτά στο Collège de και μπορείτε να συμβάλλεται απαντώντας σε αυτό το ερωτηματολόγιο ε, στην, ε, στο όλο εγχείρημα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα. Είχαμε την συζήτησή μας πάνω ε, στην έκθεση του κυρίου Σερκάς. Δεν βλέπω τους δύο πρωταγωνιστές, τον κύριο Λαμπέρ κυρίως. De Madame Edith Bauer, la discussion ε, και την συναδελφό του. Έχω εδώ έναν πάρα πολύ σημαντικό αριθμό τροπολογιών και πολύ λίγες συμβιβαστικέ προτάσεις που έχουν γίνει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εκπλήξεις στις διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες καμιά φορά. Σας δίνω λοιπόν τον λόγο για να μας ε, ε, δώσετε τις, τροπο... τις συμβαστικές προτάσεις που έχουν γίνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι δεν καταφέραμε στην ουσία να βρούμε πάρα πολλές συμβαστικές λύσεις οι οποίες να υποστηριχτούν γενικά. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία υπήρξαν συμβαστικές λύσεις, αλλά υπάρχουν και θέματα που είναι ανοιχτά. Πρέπει να περιμένουμε στην τελική ψηφοφορία για να δούμε κατά πόσο ναι ή όχι θα υπάρξει συνένεση γύρω από αυτά τα θέματα. Στην αρχή του καταλόγου ψηφοφοριών υπάρχουν τέσσερα ή πέντε θέματα όπου δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση. Είναι πολύ πιθανό θα γίνουν δεκτές δύο τροπολογίες, ενώ άλλες δύο δεν θα γίνουν δεκτές. Υπάρχουν λοιπόν θέματα όπου δεν μπορούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που καλύπτουν όλους. Και στο τέλος του καταλόγου υπάρχει ένα θέμα το οποίο αξίζει να το διεξέλθουμε. Εγώ δεν μπόρεσα ούτε και εκεί να βρω μια λύση η οποία θα μπορούσε να καλύψει όλους τους συναδέλφους. Εδώ πρόκειται ...108, 109, 103, 110, 12, 13. Για όλες αυτές τις τροπολογίες λέει η κυρία Μπάουερ. Υπάρχει κάποια δυσκολία, γιατί η κάθε τροπολογία έχει τη δική της λογική. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε αυτή την έκθεση χωρίς να λάβουμε υπόψη τον κανονισμό 561. Και υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ της οδηγίας που εξετάζουμε σήμερα και το, του κανονισμού 561 του 2006. Και γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές ο πειρασμός να ακολουθήσουμε την τακτική της χαλκομανίας στην οδηγία μας και να αντιγράψουμε κατά γράμμα τον κανονισμό 561. Αλλά στον τομέα του ελέγχου δεν θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του ελέγχου που να είναι ταυτόσιμες. Για ποιους λόγους, για λόγους οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Πρώτα απ' όλα. Διότι σε ό,τι αφορά την ρύθμιση του χρόνου εργασίας, υπάρχει μια πλειάδα διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση, μια μοναδική λύση, η οποία θα εξισφάλιζε ένα γενικό έλεγχο σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν λοιπόν ορισμένε προτάσει τροποποίηση, οι οποίε εστόχευαν ακριβώ στο να προσαρμοστεί ο κανονισμό 561 στις νέε αυτές καταστάσεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό, διότι η Εθνική Νομοθεσία έχει ήδη θεσπιστεί βάσει του κανονισμού αυτού. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία τροπολογιών, Υπάρχει μια δεύτερη σειρά τροπολογιών, που σα είπα, που μπορεί να γίνουν αποδεκτέ σε ό,τι αφορά την, τη συνέχεια πρέπει να δοθούμε, τον έλεγχο και τι ενδεχόμενε κυρώσει. Γιατί αυτέ οι τροπολογίε προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη διατύπωση του 561 και να εφαρμόσουν αυτά τα στοιχεία στην οδηγία του 2002. Αυτό όμως θα προϋπέθεται την θέσπιση ενός συστήματος το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα πολυδάπανο και θα έπρεπε να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να τα υποστηρίξω όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν κάνει κάποιες προσπάθειες για συμβαστικές λύσεις. που βασίζονται και πάλι στον κανονισμό 561 και πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν την καταγραφή από ψηφιακό ταχογράφο του χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης και εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε μια συμβαστική λύση και με τον τρόπο αυτό έχει διατυπωθεί η τροπολογία υπαριθμών 1. Σε πρακτικό επίπεδο τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα ελέγχου και τον περίφημο κανονισμό 561, η τροπολογία υπαριθμών 2 αναφέρεται σε αυτό τον κανονισμό. Είναι απόλυτα ορθό κατά την άποψή μου να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στο επίπεδο αυτό. Και εγώ έλαβα υπόψη μου τις προτάσεις των συναδέλφων μου για μια ακόμα φορά. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε μια συμβαστική λύση για την συμπερίληψη ή για την μη συμπερίληψη των ανεξαρτήτων οδηγών. Δεν μπορέσαμε να βρούμε μια λύση η οποία θα ρυθμίσει οριστικά το θέμα αυτό. Γιατί δεν μπορούμε σε ορισμένε περιπτώσει να δεχόμαστε μια τροπολογία και σε άλλε περιπτώσει να μην την δεχόμαστε σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό αυτών των οδηγών. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει την ψηφοφορία αλλά έχουμε ακόμα ένα μήνα πριν από την τελική ψηφοφορία και ενδεχομένω υπάρχει ακόμα δυνατότητα μεταξύ μας να βρούμε συμβιβαστικέ λύσεις, τουλάχιστον μπορούμε να τις αναζητήσουμε, να βρούμε νέες διατυπώσεις, να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Μπορούμε να εξευγενήσουμε ακόμα περισσότερο τις διατυπώσεις λοιπόν στο έγγραφό μας, ώστε να μην υπερφορτώσουμε την μαούνα, όπως λένε στη χώρα μου, και να μην δυσκολεύσουμε το έργο των ανεξαρτήτων εργαζομένων και εργοδοτών. Και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το έργο που έχουν φέρει σε πέρας, γιατί είχαμε 99 παραλίγο 100 τροπολογίες. Εγώ σας προτείνω να μην ξαναρχίσουμε πάλι τη συζήτηση επί της ουσίας όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, γιατί δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ο στόχο μα είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες τροπολογίες συμβιβασμού από αυτές οι οποίες μέχρι στιγμή έχουν κατατεθεί από την εισηγήτρια. Ο Στέφεν Hughes έχει το λόγο τώρα. Madam Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ Είμαι έτοιμος να συναντηθούμε όποτε θέλει η κυρία Μπάουερ για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά που προτείνει. Καταλαβαίνω το πρόβλημά της. Ε, υπάρχουν διαφορετικές θέσεις που αντανακλώνται σε, αυτούς, σε, αυτούς, σε αυτές τις τροπολογίες. Μερικές φορές οι διαφορές είναι μεγάλες, μερικέ φορές είναι μικρές. Υπάρχουν δύο διαφορετικέ λογικέ. Μερικέ φορέ να συμπεριληφθούν οι αυτοπασχολούμενοι και μερικέ φορέ να αποκλειστούν. Ε, υπάρχει μεγάλο ρήγμα εδώ και επομένω ε, δεν μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό το θέμα μέσα σε ένα μήνα όπου θα γίνει η ψηφοφορία. Κάπως βέβαια θα πρέπει να επιληθεί. Υπάρχουν και άλλε τροπολογίε που δεν έχει αναφέρει η συγγήτρια. Ε, Παραδείγματος χάρη αυτοί που αφορούν α, τους οδηγούς ε, που οδηγούν ε, φορτηγά ε, κάτω από 3,5 τόνους. Δεν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας που να τους καλύπτουν. Είναι ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το δούμε. Ίσως δεν αφορά... Δεν έχει σχέση με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συμπεριλάβουμε και τους οδηγούς αυτών των φορτηγών. Αλλιώς υπάρχει πραγματικά πρόβλημα για την ασφάλεια και την οδική ασφάλεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να περιμένουμε όμως να δούμε πώς θα αποφασίσει η Επιτροπή για αυτό το κρίσιμο σημείο της συμπερίληψης ή αποκλεισμού των αυτοαπασχολούμενων. Και ελπίζω να επιληθεί αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνάδελφος. κυρία Τιούρενεν. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε μόνο δύο συμβαστικές τροπολογίες επιτάπητος. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν για την εφαρμογή και τον έλεγχο νομίζω. Πολλοί βουλευτές από ανεξάρτητα από την πολιτική του ομάδα θέλουν να εξασφαλίσουμε, ας ευχαριστώ για τον καφέ, ότι θα έχουμε τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικά μέτρα, τα οποία όμως θα εφαρμόζονται και θα ελέγχονται στα κράτη-μέλη. Γιατί αλλιώς καλή είναι η νομοθεσία, αλλά αν δεν εφαρμόζεται τι νόημα έχει. Υπάρχουν λοιπόν ίσως περισσότερες δυνατότητες ε, για να το καταφέρουμε αυτό. Αλλιώς, τι άλλο να σας πω. Μία μόνο τροπολογία έχουμε καταθέσει, σαφή. Ε, είναι μια θέση αρχής για την διαδικασία που έχει επιλεγεί, αλλά και για το περιεχόμενο. Γι' αυτό έχω ε, υποβάλει μετροπολογία τροπολογία για να αρνηθούμε την πρόταση της Επιτροπής. Κύριε Πάουερ, ίσως δεν είναι αυτή μια πρόσκληση συμβιβασμού. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις προκειμένου να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάποια πράγματα για την εφαρμογή των έλεγχων. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Φιγκερέιδο. Ε, ε, ε, Συγγνώμη, έχω δυσκολίες κατανόησης για αυτή την συμβιβαστική πρόταση. Διότι δεν μπορώ να κατανοήσω σε τελική ανάλυση πώς στην πράξη θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των ανεξαρτήτων εργαζομένων όταν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Αν υπάρχει λοιπόν μια νομοθεσία η οποία θα είναι αυτόσιμη, ταυτόσιμη για όλους, θα ήθελα να κατανοήσω λίγο καλύτερα ποια είναι η άποψη της κυρίας Μπάουερ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν, δεν θέλετε να μιλήσετε. Α, θέλετε βέβαια. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την κυρία Μπάουερ. Πήγε όσο μακριά μπορούσε μάλλον για να εξεύρει τους ε, συμβιβασμού. Μερικές φορές δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποιο όριο στου στους Έκανε ό,τι μπορούσε. Τους υποστηρίζω τους συμβιβασμού αυτούς, αλλά συμφωνώ ότι είναι αμάλλον αδύνατο να βρούμε μία λύση για αυτό το θέμα. Ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε τελικά. Αλλά καταλαβαίνω και υποστηρίζω τη δουλειά της κυρίας Μπάουερ. Pas nécessaire. κανείς όχι, κυρία Μπάουερ, για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση για τους δύο συμβασμούς. Ακούσατε τις αντιδράσεις των συναδέλφων και τη διάθεσή τους να κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουμε λιγάκι, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο εφαρμογής και τα μέσα εφαρμογής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. ο Στέφαν Χιούς ε, εξήγησε και περιέγραψε ανάγλυφα την κατάσταση. Υπάρχουν δύο τάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες. Είναι δύσκολο να τις συγκεράσουμε τις τροπολογίες αυτές. Έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα το καταδύναμεν. Και φυσικά θα κάνω πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορώ για να βρω και άλλες λύσεις στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Είμαι έτοιμη να συναντηθούμε με τον κύριο Χιούς. Έχουμε βρεθεί ούτω ή άλλω ήδη και τα έχουμε πει και κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά χρήσιμη και βαθιά για την πρόταση. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων, αν διατηρηθεί αυτή η πρόταση, νομίζω ότι αυτό είναι το όριο. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις ότι θα πρέπει να κατέβουμε από το, τους 3,5 τόνους. Άλλες προτάσεις λένε ότι θα πρέπει να υπερβούμε τους 3,5 τόνους. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Ε, εγώ νομίζω δεν μπορούμε να πάρουμε υπόψη όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τα οχήματα 3,5 τόνων. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το έργο της, α, του χτενίσματος, αν θέλετε, των νομοθετημάτων στην Επιτροπή Μεταφορών. Αυτή θα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό. Έχουμε και την πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών για το θέμα αυτό. Το κείμενο που έχουμε ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει εγκριθεί ποτέ. Και έτσι διαφαίνεται πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, γιατί η ίδια η Επιτροπή Μεταφορών τελικά δεν έχει οθετήσει καμία γνωμοδότηση. Συνέταξε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει οθετηθεί όμω. Πρόεδρο, για το θέμα αυτό θα ψηφίσουμε στην συνεδρία του Απριλίου, 28 Απριλίου, και μέχρι τότε θα δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε τη σύγκληση με την εισηγήτρια. Έχουμε πέντε λεπτά πριν από την ψηφοφορία. Δυστυχώς η κυρία Λαομπέρ και η κυρία Πικεβισούτετς που μου είχαν πει ότι θα ήταν εδώ το πρωί, δεν είναι εδώ. Ας δώσω το λόγο στον κύριο Σέρκας για να κλείσουμε τη χθεσινή συζήτηση. Α, δεν σας ξέχασα. Ξέρω ότι η Επιτροπή είναι παρούσα και θέλει να αναφέρει τη δική της άποψη. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον κύριο Ολιβιέ Τέλ, για να μας πει την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ε, θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέρκα για το σχέδιο χνομοδότησης. Ε, συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή, ε, δηλαδή ότι η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση όχι μόνο είναι ευκταία, αλλά είναι και δυνατή. Εφόσον ε, πετύχουμε τους κατάλληλους συμβιβασμούς. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό για την ε, ισότητα της μεταχείρισης. Χθες ε, διαρωτηθήκαμε για την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Διαρωτηθήκατε. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει δυσκολία για την ε, τροπολογία 12 που είναι πολύ σημαντική για τον εισηγητή και για όλους μας τελικά. Για την 8 και 4 θεωρούμε ότι οι τεχνικές λύσεις επίσης είναι δυνατές το θέμα το πιο δύσκολο είναι η τροπολογία 13 για το θέμα των δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας πω για αυτό το θέμα ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι ακριβώς αυτή που θα ήθελε ο εισηγητής μας, τα είπα αυτά. Απλώς η... πρέπει να πούμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και σε σχέση με αυτή την κατάσταση η πρόταση της Κομισιόν σηματοδοτεί κάποια πρόοδο και εγγυήσεις για τους μετανάστες εργαζόμενους. Είναι καλύτερη λοιπόν η πρόταση, είναι και καρπός συμβιβασμού ανάμεσα στην ε, διάθεση για να υπάρξει ίση μεταχείριση και την ανάγκη όμως να λάβουμε υπόψη κάποιους δημοσιονομικούς, οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη και υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Τώρα, η λύση για αυτό το πρόβλημα προφανώς είναι δύσκολη και περίπλοκη, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη τα δικαιώματα ε, βασίζονται στις συνεισφορές, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη ε, βασίζονται στην κατοικία. Κάποια κράτη-μέλη, ακόμα και με τον ε, σημερινό περιορισμό, μας λένε ότι ήδη το έχουμε, πάει υπερβολικά μακριά. Και όταν ε, τα δικαιώματα βασίζονται στην κατοικία, τελικά καλύπτει η πρόταση περισσότερους ανθρώπους από τους σημερινούς εργαζόμενους. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, Πρόεδρε, είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο συνομοθετών, δηλαδή Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Έχουμε λάβει την εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξαναδούμε την κατάσταση μέχρι το 2013-2014. Ε, σήμερα Βέβαια, και το λέει η οδηγία, τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που λέει το κείμενο. Θα μπορούσαμε να ξαναδούμε την κατάσταση λοιπόν ε, στο μέλλον για να βελτιώσουμε τα πράγματα και να παγιοποιήσουμε τα δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερ, η κυρία Ελκεβισούδε δεν έχουν έρθει ακόμα ο κύριος Σέρκας. Las últimas palabras del representante de la Comisión. Θέλω ευχαριστήσω αυτά που είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να προχωρήσουμε στι τροπολογίε 4, 8 και 12, που είναι πάρα πολύ σημαντικέ και δεν χάνω την, ευκαι... την ελπίδα ότι η τροπολογία παριθμό 13 θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τι επόμενε μέρε. Όπω είπα χθε και όπω επαναλαμβάνω σήμερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα για να να καταλάβω τι δυσκολίε που μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένα κράτη-μέλη ή τι δυσκολίε που μπορούν να δουν στην τροπολογία τη δική μου για τα ωφέλη αυτά τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν προς τους μετανάστες εργαζόμενους πέραν αυτών που απορρέουν από την μόνιμη κατοικία ενός εργαζόμενου, όπως αναφέρεται στην νομοθεσία. Ο στόχος μου δεν είναι να διευρύνω αυτά τα δικαιώματα είτε να παραβιάσω την αρχή τη επικουρικότητα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε χώρα χωριστά τα θέματα αυτά. Δηλαδή δεν πρόκειται να θίξω τα εθνικά συστήματα κοινωνική ασφάλιση και τη φιλοσοφία που τα διατρέχει. Το μόνο το οποίο θέλω να επιτύχω είναι να εδρεωθεί η αρχή τη μη διάκριση συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων όπου υπάρχουν λύσεις για αυτά τα θέματα σε άλλους κώδικες, σε, άλλους οδη... σε άλλες οδηγίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε διατυπώσεις που να λένε ότι το θέμα αυτό θα επιληθεί οριστικά σε άλλα νομικά εργαλεία, σε άλλα νομοθετήματα. Είναι δυνατότητες που θα μπορέσουμε να τις μελετήσουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω και το κάνω για να απαντήσω στην κυρία Όιμεν Ρόιτεν και την άλλη συνάδελφο η οποία έλαβε τον λόγο χθες ότι σε αυτή την οδηγία, όπως μας είπε και η ίδια Κομισιόν στο εγγραφό τη, δεν εκχωρούνται ή τροποποιούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία παραμένουν μέσα στην εθνική κυριαρχία. Αυτό το οποίο λέει σε η οδηγία αυτή είναι ότι όποιος μένει και εργάζεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με ένα ηθαγενή εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται σε ίσες, σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ισότητα μεταχείρισης και μόνο να έρεται αυτό όταν υπάρχει η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την ε, διαδικασία σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας. Ξέρω ότι η Κομισιόν κάνει κάτι θετικό όταν αναφέρεται στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά σε περιπτώσεις που έχει να κάνει με οικογενειακά επιδόματα και με ε, διάφορες, ε, διάφορα ωφελήματα τα οποία μπορεί να έχει ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας του, αυτό δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζομένου και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω καμία αιτιολόγηση στην στάση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί σωστά. Πρέπει ή να το ρυθμίσουμε τώρα ή να πούμε στο, στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη θα επιληθεί το θέμα αυτό σε μεταγερέστερες οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ας σταματήσουμε εδώ προς το παρόν για το θέμα αυτό. Και στην επόμενη φάση θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών καταρχήν που τρέχει μέχρι τις 24 Μαρτίου, όπως συμφώνησε και ο εισηγητής, και πέραν της 24 Μαρτίου θα γίνει μια συζήτηση για τις τροπολογίες που θα έχουν κατατεθεί μέχρι τότε. Δεν το έχω αυτό στα χαρτιά μου και άμα δεν το έχω στα χαρτιά μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, λέει ο πρόεδρος. θα κάνουμε μια συζήτηση στις 27 Απριλίου και θα ψηφίσουμε στις 28. Δεν είναι ιδανικού χαρακτήρα αυτή η ρύθμιση, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ξεκινώντας με το σημείο 11, όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Μπαστός για το Περιφερειακό Ταμείο. Κυρία Μπάστος, σας είπα ότι μίλησα με την κυρία Ντανούτα Χιούπνερ χθε και τη είπα ότι μέσα στα πλαίσια ενό πνεύματο αγαστή συνεργασία των δύο επιτροπών μα είναι απαραίτητο να μπορέσει να λάβει υπόψη τις τροπολογίε που εμεί θα εγκρίνουμε επί τη βάση τη γνωμοδότησή σα, δεδομένου του ότι δεν θα θίξουμε ορισμένα σημεία κέριου χαρακτήρα τα οποία θα δυσκολέψουν τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτή την διευκρίνηση θα γίνει αποδεκτή και η άποψη της Επιτροπής μας όπως εκφράζεται με τη γνωμοδότηση. Άρθρο 1, 4, σημείο 1, τροπολογία 15, σούτερ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Απορρίπτεται. 16 κόσα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17 κρέτσου ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται πρέπει να ελέγξουμε. Ψήφι υπέρ και πάλι. Με, με ηλεκτρονικό τρόπο. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας. Όχι, κυρία Φιγερέδο δεν την έχει, αλλά εμείς θα την καταμετρήσουμε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Περιμένουμε την πρώτη αντιπρόεδρο, μήπως ψηφίσει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 19 υπέρ 13 κατά, γίνεται δεκτή. Επομένως, τροπολογία 18 της κυρίας Κρέτσου. Κύριε Χάντελ, και εσείς δεν έχετε την κάρτα σας. Καλά, δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Κυρία Κρέτσου, έχετε την τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Πόχες. Το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. 19 Σρόντερ, ψήφι υπέρ. Κατά. Θα έλεξουμε ηλεκτρονικά. 19. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Κυρία Φιγκερέτου, κατά τη στάση αποχής, εντάξει. Ψηφίσαν όλοι, μάλιστα. Πέρας. 21 ψήφοι κατά 11 υπέρ απορρίπτεται σαφώς. Κύριε Κλάρκ, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, είμαι άκαρτος. Θα μου εξηγείτε λοιπόν ποια είναι η θέση σε κάθε ψηφοφορία. Τροπολογία 20 Σρέντερ λοιπόν, την ψηφίσαμε όμως αυτή νομίζω ή όχι. 20 την ψηφίσουμε υπέρ κατά απορρίπτεται, ναι. 4 της εισηγήτριας για διαγραφή ψήφι πέρ, κατά αποχές δεκτή, 29 της κυρίας Ζίπελ, ψήφι πέρ κατά αποχές δεκτή. 22 και 23 είναι ταυτόσιμες, ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτές. 24-25 επίση είναι ταυτόσιμες, ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτές. 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Μετά την αιτιολογική σκέψη 2, τροπολογία 9 με προφορική τροποποίηση, ψήφι υπέρ της 9 όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ κατά δεκτή. Μετά την αιτιολογική σκέψη 1, τροπολογία 5 της κυρίας Γκιόντς, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στη συνέχεια Τροπολογία 6 για την αιτιολογική σκέψη 2 της κυρίας Γκούνς, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 της κυρίας Ζίπελ, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8 της κυρίας Πιτσότο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή η ένα εκπίπτει, περνάμε στην τροπολογία 10 της κυρίας Μπιτσότο, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, Δύο της Ήτριας, ψήφι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 12 της κυρίας Μεσνέρ, ψήφι κατά αποχές δεκτή. 3 της εισηγήτριας, εκπίπτη 11 της κυρίας Ζίπελ, ψήφι κατά αποχές δεκτή. 13 της κυρίας Ζίπελ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 εκπίπτη όχι, όχι, δεν εκπίπτει. Ψηφίζουμε τη 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κυρία Κλάρκ, τι λέτε. Κατά. Κατά, μάλιστα. Δύο ψήφοι κατά, λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 32 ψήφοι υπέρ, Δύο κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η γνωμοδότηση. Συγχαίρουμε την κυρία Μπάστος. Alors, nous venons à de Γνωμοδότηση Κρίστενσεν στο σημείο 12 για τις ανάγκες ιδίων πόρων σε ό,τι αφορά την ε, προληπτική εποπτεία σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αποδοχών. Άρθρο 1, τροπολογία 14 του εισηγητή, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 του ιδίου υπέρ. I will take the TER now. 17 euh, du rapporteur qui est pour. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 του ιδίου, του εισηγητή δηλαδή 18 υπέρ. Κύριε Ελμέ. Κυρία Πρόεδρε, από ό,τι λέω, μιλάτε πολύ γρήγορα και λέτε ότι εγκρίθηκε κατευθείαν. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Άκουσα ποιος είναι υπέρ, εγκρίθηκε. Αυτό άκουσα εγώ. Ωραία, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, διορθώνω. 18 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ωραία κύριε Έλμερ, εγκρίνεται. Τόμας Μαν, 53, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 του εισηγητή, ε, καταπίπτει, 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 22 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 του κυρίου Λεγιαρίκ και της κυρίας Τσίμερ υπέρ 55 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 του κυρίου Ιαρίκ και Τσιμέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 του εισηγητή καταπίπτει περνάμε στην 57 υπέρ παρακαλώ κατά Α, ξανά την 57 παρακαλώ θα κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό έχετε κάρτα κύριε Κλάς Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 24 υπέρ. Λάθος, διορθώνει η πρόεδρος. 25 υπέρ και 13 κατά. Εγκρίνεται άρα η τροπολογία. Περνάμε στην 25 εισηγή του υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 58 Υπέρ παρακαλώ της κυρίας Δέλη. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 του κυρίου Λεγιαρίκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 του εισηγητού Εκπίπτει 27 και περνάμε στην 28 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61. Ψηφίζουμε του κυρίου Λεγιαρή κυρία Τσίμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 της κυρίας Δελή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 της κυρίας Δελή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές ένα λεπτό θα επαληθεύσουμε, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, 31, άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Κλάρκ, πώ ψηφίζετε. Είστε κατά υπέρ. «29 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, οπότε εγκρίνεται» δεν είχα δει καλά δηλαδή. 64 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 της κυρίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην 32 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 της κυρίας Δελή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην τροπολογία 33 υπάρχει μια προφορική τροπολογία η οποία προτάθηκε η οποία δίνει μία νέα εκδοχή όπου διορθώνεται η λέξη should ε, και στη θέση της λέξης shall, θα έπρεπε και όχι πρέπει. Λοιπόν, υπάρχει αντίθεση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι, λοιπόν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 του εισηγητή, υπέρ, κατά, Αποχές ε, παληθεύουμε ηλεκτρονικά. Εψήφισαν όλοι πέρας. 20 ψήφοι υπέρ και 18 κατά. Οπότε η τροπολογία 35 εγκρίνεται. Η 67 τώρα της κυρίας υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 36 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 πάλι του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 του ιδίου υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. κύριος Σκάκη και η κυρία Φιγκερέντο ψηφίζουν επίσης. Οπότε έχουμε 20 υπέρ, 18 ψήφους κατά, άρα εγκρίνεται. 68 της κυρίας Δελή καταπίπτει. Το ένα του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δύο του εισηγητή είναι ταυτόσιμη με την 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, τρία του εισηγητή υπέρ κατά Τώρα ερχόμαστε στη συμβιβαστική τροπολογία που κατατίθεται από τέσσερις ομάδες, πέντε μάλλον. Υπάρχει και μια προφορική τροπολογία, σας υπενθυμίζω, η οποία επίσης κατατέθηκε. Σας τη διαβάζω. Committees as part of their governance structure, full stop, and then remuneration committees will go on. Il n'y a pas d'opposition cet amendement. Υπάρχει αντίθεση σε αυτή την τροπολογία. Όχι, οπότε ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται ε, καταπίπτουν όλες οι άλλες τροπολογίες. Στο 5 της αιτιολογικής σκέψης έχουμε τη 44, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 του Τόμας Μαν με μια προφορική τροπολογία η οποία ζητά την προσθήκη στο τέλος του κειμένου Δεν ξέρουμε τι είναι το EFQM, λέει η πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Ναι, ο εισηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Θα πρέπει να μιλάμε για το υπόδειγμα μετά το EFQM. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο. Το M δεν σημαίνει model στο EFQM. Μήπως πρέπει να γράψουμε απλώς EFQM ολογράφος. Και μετά να βάλουμε και εισαγωγικά μετά το EFQM θα είναι σαφέστερο για όλους. Κύριε Έλμερ, διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να εξετάσουμε μια προφορική τροπολογία, μήπως μπορεί να μας εξηγήσει καν, κάποιος τι σημαίνει αυτή η ακροστοιχίδα. Όλη η αλήθεια να λάμψει για το EFQM λέει η Πρόεδρος πρέπει. ένα υπόδειγμα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δείτε τα θέματα της ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αφορά την, ε, το σχεδιασμό στόχων κτλ. Το ερώτημα όμως είναι, κύριε Άλμερ, μια στιγμή, χαλαρώστε. Και εγώ ανησυχώ όπως και εσείς. Το M το καταλάβαμε, είναι το μόντελ. Το ε είναι equivalent. Equivalent, fair, ισοδύναμη, δίκαια λοιπά. Λοιπόν, μια στιγμή θα το βρω. European Foundation for Quality Management Model. Μπράβο. Είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την ποιότητα της διαχείρισης, το μοντέλο της Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη διαχείριση της ποιότητα. Καταλάβαμε τι σημαίναν αυτά τα κορακίστικα σε αυτή την τροπολογία που αν δεν υπήρχε καμία αντίδραση θα την είχαμε εγκρίνει ούτω ή άλλω. Μπορείτε λοιπόν να συμπληρώσετε την τροπολογία με εκπεφασμένη μνήμα όλων αυτών των στοιχείων τη ακροστοιχίδα. Ποιο είναι υπέρ λοιπόν τη τροπολογία, κύριε Μάν, μετά από όλα αυτά. Κατά. Αποχε. Εγκρίνεται με το EFQM και το μοντέλο από πίσω. Η 5 του εισηγητή εκπίπτει και έχουμε τη 46 η οποία επίσης εκπίπτει και μετά περνάμε στη αιτιολογική σκέψη 5 και έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση Β από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχέσα. απορρίπτεται. θα δούμε, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το Β. Υπάρχει μια... Ε, πώς ψηφίζετε κύριε Κάτ, κύριε Φιγκερέντο, υπέρ, ωραία. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι, πέρας. Έχουμε 15 ψήφους υπέρ και 23 ψήφους κατά, άρα απορρίπτεται. Στη συνέχεια 47 που ζητά ένα νέο σημείο στην αιτιολογική σκέψη. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 48 της κυρίας Δελή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά έχουμε την τροπολογία 7 του συγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στο, στην αιτιολογική σκέψη ε, ε, όχι εδώ λέει, διορθώνει η πρόεδρος. Έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση υπέρ κατά αποχές, η σε εγκρίνεται ε, και ερχόμαστε στις 49 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε μια συμβαστική τροπολογία D. Πέντε ομάδες την προτείνουν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στο έξι της αιτιολογικής σκέψης η 10 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 του εισηγητή πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 12 της αιτιολογικής σκέψης έχουμε την συμβαστική πρόταση ε υπέρ κατά αποχές. Μετά είναι η τροπολογία 13 του εισηγητή υπέρ κατά υπέρ λέω κατά εγκρίνεται Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. και κάτω. Ψήφισαν όλοι πέρας. 35 υπέρ, 4 ψήφοι κατά, 0 αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Κρίστενσεν. Στη συνέχεια έχουμε ψηφοφορία της γνωμοδότησης του κυρίου Λογιαρίκ Στην παραγράφο 1 έχω την τροπολογία τη συμβιβαστική παρουσιάζουν τέσσερις ομάδες Β. Υπέρ. Θα έπρεπε πριν να αρχίσω την ψηφοφορία να το είχατε δηλώσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Διαδικαστικό. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η συμβιβαστική πρόταση και οι άλλες. Είχαμε μόνο τα γαλλικά, ήρθαν πάρα πολύ αργά στα χέρια μας, οπότε δεν μπορέσαμε ούτε καν να τις ε, διαβάσουμε, να τις εξετάσουμε και δεν ξέρουμε πάνω σε τι κείμενο ψηφίζουμε. Ωραία, το σημειώνουμε. Στην παράγραφο 2, συμβαστική τροπολογία σε, που παρουσιάζεται από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά 16 του κυρίου Κοφεράτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 του ιδίου ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Madame Figueredo, c'est pas d'une originalité folle ce matin. Alors. Εψήφισαν όλοι. Ε, η κυρία Μόρα, νομίζω κάνατε λάθος. Κατάλαβα, λέει η πρόεδρος. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Έχουμε 18 ψήφους υπέρ, 22 κατά. Οπότε απορρίπτεται την τροπολογία του κυρίου Κοφεράτη στην παράγραφο 3. Έχω την συμβαστική 2 που παρουσιάζεται από τέσσερις ομάδες. Ψήφι παρουσιάζεται είπα από τέσσερις ομάδες ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και στη συνέχεια έχουμε την τροπολογία 11 της κυρίας Δέλη όπου έχει ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία Το τρίτο μέρος της τροπολογίας ε, ε, θα ψηφιστεί γιατί είναι αυτό το τρίτο μέρος σύμβατο με την συμβιβαστική λύση που προτείνεται. Συμβαστική λύση D. Θα βρω το κείμενο και θα σας το διαβάσω λέει η Πρόεδρος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 στις επιχειρήσεις όπου έχουν, υπάρχουν θυγατρικές ε, ζητά να υπάρξει λειτουργία της απαγόρευσης της, των κρατικών βοηθειών ή των βοηθειών που προέρχονται από την ΕΕ. Ποιος είναι λοιπόν υπέρ αυτής της, ε, του τρίτου μέρους της ε, συμβιβαστικής πρότασης της τροπολογίας της κυρίας Δελή. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Η 11 απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 3 έχουμε την ε συμβιβαστική. Τέσσερις ομάδες την προτείνουν. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 27 υπέρ. 20, ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 4, τροπολογία 29, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 συμβατή με την προηγούμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά 32 της κυρίας Δελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 6, τροπολογία 33, που είναι τροπολογία που ζητεί κατάργηση. Ψήφι υπέρ παρακαλώ, μεγάλη κατάργηση, υπέρ, ε, κατά. Ας επαληθεύσουμε εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Κλάκ, πώς ψηφίζετε, κυρία Φιγκερέιντο, είστε κατά και οι δύο, ωραία. Λοιπόν, Πέρα της ψηφοφορίας 23 υπέρ, 17 κατά, οπότε εγκρίνεται η 33. Μετά από την παράγραφο 6, η παράγραφος 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7.37 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. η 38 είναι συμβατή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 39 παράγραφος 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 40 του κυρίου Κοφεράτη υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 41 Μπαλτασάρ και Μεσνέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9.42 των ιδίων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 ρενιέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 τελεί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 σογκόρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 1 και 2 μαζί τα βλέπουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική τροπολογία στο Β που κατατίθεται από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ερχόμαστε τώρα στην, στο, δύο, στο Β της αιτιολογικής σκέψης και Έχουμε εδώ την 8 κυρία Σιμπέλ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 9 είναι συμβατή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στο ε της αιτιολογικής σκέψης τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης ψηφίζουμε ηλεκτρονικά κύριε Κλάρκ, υπέρ, κύριε Φιγκερέντο, και η κυρία Μωρά. Ψήφισαν όλοι. Εψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Έχουμε 31 ψήφους υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές, οπότε συγχαρητήρια στον εισηγητή εγκρίθηκε. Ερχόμαστε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία της πρωινής μας συνεδρίασης τη γνωμοδότηση του κυρίου Σέρζιο Κοφεράτη Στην παράγραφο 1 έχουμε μια τροπολογία συμβιβαστική 1 που κατατίθεται τον εισήγητη ψήφι παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 1 τροπολογία 5 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Σήμερα το πρωί η ομάδα φιλελευθέρων μου ζήτησε να ψηφίσουμε χωριστά αυτή την τροπολογία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και αν μου επιτρέπετε θα σας πω πού θα κάνουμε το διαχωρισμό της τροπολογίας. Πώς θα τη χωρίσουμε. Για ποια τροπολογία μιλάτε. Το πρώτο τμήμα, πρόεδρος διακόπτη. Θέλετε χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Κατάλαβα καλά. Ε, θα σας πω τη, τη γνώμη μου για τη συνολική τροπολογία, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε χωριστά. Η Πρόεδρος, κύριε Σιγητά, μπορείτε να μας πείτε Πού θα χωρίσουμε την τροπολογία. Το πρώτο σημείο. Τελειώνει με τη φράση μέχρι το ποσοστό ανεργίας να κατέβει με τρόπο ουσιαστικό και βιώσιμο και διαρκή. Και το δεύτερο σημείο δείχνει ότι το κράτος, το κοινωνικό κτλ. κτλ. Έχω θετική γνώμη για την ε, τροπολογία συνολικά. Εγώ, εγώ την παρουσίασα εξάλλου. Ε, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα, εφόσον ε, οι φιλελεύθεροι το θέλουν, να την ψηφίσουμε χωριστά. Ωραία, λέει Πρόεδρος. Ψηφίζουμε τότε χωριστά. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας τονίζει ότι η ανάκαμψη είναι εύτραυστη και η ανεργία συνεχίζεται μέχρι, μέχρι να μειωθεί ουσιαστικά, μέχρι το σημείο, να έχει μειωθεί ουσιαστικά και με διαρκή τρόπο, υπέρ, κατά, εποχές. Υιοθετείται το πρώτο τμήμα. Τώρα πάμε στην ψηφοφορία του δεύτερου του βήματος, το υπόλοιπο του κειμένου και τονίζει μέχρι συνεισφέρει στην ανάκαμψη. Ποιος είναι υπέρ αυτού του δεύτερου τμήματος. Κατά. Υιοθετείτε και αυτό δεύτερο τμήμα. Πάμε στην τροπολογία 6 κυρία Φιγκερέ, της κυρίας Φιγκερέιδο, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 της Ιδίας, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8 με που θέλει να βάλει έναν υπότιλο. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Παράγραφος 2. Ψηφίζουμε μια τροπολογία συμβιβαστική την υπαριθμόν Β που παρουσίασε ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Πάμε στην παράγραφο 3, συμβαστική τροπολογία σε, γάμα υπέρ, κατά, αποχές, θα το επαληθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι πέρα τις ψηφοφορίες. 20 υπέρ, 18 κατά, δύο αποχές. Η συμβαστική τροπολογία σε υιοθετείται. Μετά τροπολογία 16 υπέρ, κατά, δεν σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Κύριε Κλάρκ. Ψήφισαν όλοι πέρας της 24 υπέρ, 13 κατά, 3 αποχές υιοθετείται. Παραφός 4, συμβαστική τροπολογία δέλτα υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Μετά, τροπολογία 21 του εισηγητή, παραφό 4, κατά αποχές απορρίπτεται. 22, παράφος 22. Υπότιτλος που εισάγει ο εισηγητής υπέρ κατά υιοθετείται η συμβαστική τροπολογία ε υπέρ στην 5. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 24. Είναι συμβατή. Την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 25, τροπολογία 25, κοφεράτη, υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Πράγματος 6, τροπολογία 26, φιγκερέιδο, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 27, υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Η τροπολογία 28 είναι συμβατή, την ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 29. Με Υπότιτλο που βάζει ο εισηγητή υπέρ κατά αποχέ υιοθετείται. Πράγμα 7. Συμβαστική τροπολογία F του εισηγητή υπέρ κατά αποχέ θα το επαληθεύσουμε. Κυρία Φιγκερίδα, το ψηφίζετε. Ο Κλάκ είναι κατά. Κυρία Φιγκερίδα απέχει. Πέρα ψηφοφορία. 18 ψηφί υπέρ. 19 κατά. 3 αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. λόπε. Φοντάνε. Φοντανιέ. Υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε τροπολογία 30. Όλοι ψήφισαν 23 υπέρ, 17 κατά. Τροπολογία Φοντανιέ υιοθετείται. Μου λένε ότι και οι υπόλοιπε τροπολογίε είναι συμβατέ, θα τι ψηφίσουμε. Δεν ξέρω τι θα, το τρέσμα θα βγει στο τέλο, αλλά ψηφίζουμε. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 32. Πλην. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα επαληθεύσουμε την 33. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφι υπέρ, 20 κατά, υιοθετείται με μία ψήφο υπέρ. Τροπολογία 34 κοφεράτη υπέρ για την παράγραφο 7. Κατά αποχές υιοθετείται. Παράγραφος 8. Τροπολογία 35 φιγκερέιδο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26. 36 γνώμη. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Παράγραφος 8. 37, τροπολογία 37 των ιδίων. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 38, Φιγκερέιδο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39, Λόπε Φοντανιέ υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 40, Λίνε, συμβατή. Την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ο κύριος Κλάκ είναι κατά. Η κυρία Φιγκερέιδο απέχει. Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψηφί υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Υπήρχαν και δύο εποχές. Τώρα πάμε στο σημείο 15 της σημερινής διάταξης. Θα παραδώσω την Προεδρία στην Αντιπρόεδρο κυρία Λίν για να παρουσιάσει αυτό το σημείο. Yes, Περνάμε τώρα στην ε, μελέτη. Ζητήσαμε να γίνει αυτή η μελέτη για να έχουμε και κάποιες κατευθύνσεις σε σχέση με τα θέματα της κοινωνικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της ατζέντα για τα κοινωνικά θέματα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο ε, για το, από το Ινστιτούτο για τα εργασιακά θέματα για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσοχή τους. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσω τα πορίσματα της μελέτης μας για την κοινωνική ατζέντα στο τέλος της δεκαετίας του 1990, αρχές δεκαετίας του 2000. Η μελέτη αυτή έχει γίνει μετά από αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί και με τη συνάδελφό μου την Μπάρμπαρα που είναι εδώ και τον κύριο Μάικελ Κέντζια από, επίσης από το Ινστιτούτο για τις Εργασιακές Μελέτες στη Γερμανία. Αυτό το οποίο μου είπαν η μελέτη αλλά τα, και τα κύρια πορίσματά της, οι διαφάνειες αυτές έχουν διανεμηθεί σε όλους ή διανέμονται αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλουν να φύγουν να αποχωρήσουν ησύχω και ηρέμος παρακαλώ, λέει η πρόεδρος για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση. Ευχαριστώ, συνεχίστε παρακαλώ. Νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε το περιεχόμενο αυτής της μελέτης τα, οι διαφάνειες είναι στα χέρια σας, έχουν διανεμηθεί για την αναδίδυσή σας. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα κύρια πορίσματα αυτής της μελέτης και να συζητήσουμε μαζί σας για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Πέντε βασικά σημεία. Καταρχήν το γενικό πλαίσιο της μελέτης. Θα ακολουθήσω και οι στόχοι της μελέτης, στην κατάσταση των πραγμάτων στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Θα συζητήσω μετά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος στόχος της ε, μελέτης αυτής ήταν να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλος ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ατζέντα των ετών 2000 με 2005, 2005 έως 2008 και αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε σχέση με την ε, ανανεωμένη ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα σε σχέση με τα επιτεύγματα μέχρι τώρα και να εξετάσουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο στην προώθηση αυτή τη ατζέντα για να δούμε πού βρίσκονται οι ευκαιρίε, πού βρίσκονται τα προσκόμματα για τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες από τις διαφάνειες οι οποίες είναι διανεμημένες, να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση των κυρίων εξελίξεων τις οποίες ερευνήσαμε εμείς από το τέλος της δεκαετίας του 1990 αρχές της δεκαετίας του 2000, μια χρονική περίοδο όπου ξεκίνησε η διαδικασία <clears throat> οικοδόμησης μιας πολιτικής επί τη βάση ήδη προηγουμένως υφιστάμενης νομοθεσίας και επί του λεγόμενου ήπιου νόμου που βασιζόταν στη διαδικασία της ε, Λισαβόνας. Έκτοτε έχει μειωθεί το κομμάτι το οποίο έχει ε, νομοθετικό χαρακτήρα, αλλά αντίστοιχα διευρύνθηκε το φάσμα των πολιτικών μέχρι σήμερα. Η έκθεσή μας περιλαμβάνει λοιπόν πάρα πολύ λεπτομερείς περιγραφές των πρωτοβουλειών σε νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υπείου νόμου που εγκρίθηκαν μετά από το 2000 επί τη βάση της στρατηγικής Λισαβόνας και επίσης το 2008 μπορούμε σε όλα αυτά να διακρίνουμε μια έντονη φάση νομοθετικής δραστηριότητα, ιδιαίτερα από το 2000 ως το 2005 με πέντε κυρίες προτεραιότητες καταρχήν την προετοιμασία της ενδιάμεσης ε, μετα... ε, αναθεώρησης της στρατηγικής Λισαβόνας, πλήρη απασχόληση και ποιότητα εργασία, ποιότητα κοινωνικών πολιτικών, ποιότητα εργασιακών σχέσεων, διεύρυνση και διεθνή συνεργασία. Εγώ βασίστηκα, όλοι βασίστηκαμε στην έκθεσή μας αυτή, σε ανταλλαγές απόψεων και συνεντεύξεις, αλλά επίσης αναλύσαμε και την κοινωνική πολιτική και την νομοθεσία για τα έτη μετά το 2007, όπου υπήρχε αυξανόμενη ετερογένεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δυσκόλεψε την πρόοδο σε νομοθετικά θέματα και μπορούσαμε να δούμε και την ε, αυξανόμενη επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κέρια νομοθετικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Τώρα, αν έρθουμε σε πιο πρόσφατα ζητήματα, η ανανεωμένη στρατηγική της Κομισιόν για τα κοινωνικά θέματα του 2005 δημιούργησε ένα ευρύτερο χώρο παρέμβασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στην κοινωνική πραγματικότητα και επειδή διευρύνθηκε και ο τομέας ο οποίος καλύπτεται από τις νομοθετικές δραστηριότητες, αλλά επίσης και από τον ήπιο νόμο, μέσα σε εισαγωγικά. Υπάρχουν λοιπόν μερικέ προοπτικέ οι οποίε ξεκίνησαν, οι οποίε δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρω. Το πρώτο τμήμα τη μελέτη μα λοιπόν κλείνει με μία αποτίμηση αυτών που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 10 με 15 χρόνια και αυτό το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι έχει τροχοπεδηθεί η νομοθετική δραστηριότητα από την ετερογένεια απόψεων στο Συμβούλιο, ιδίως μετά από την διεύνηση, όταν η σύνθεση του Συμβουλίου έχει προφανώς τροποποιηθεί και αποτελεί αντικείμενο, αποτελεί εμπόδιο για την έγκριση νέων νομοθετημάτων και πολλοί θέλουν να διατηρήσουν το status quo σε σχέση με τις εργασιακές ρυθμίσεις, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το τροποποιήσουμε τώρα. Αυτό δείχνει ότι κάποια ζητήματα είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν και βλέπουμε αυτές τις δυσκολίες για την οδηγία για το χρόνο εργασίας ή επίσης για την, στα πλαίσια της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Είναι δύσκολο λοιπόν να προωθήσει κανείς είτε στο Συμβούλιο είτε στην ε, Κομισιόν δραστηριότητες προς τον τομέα αυτό. Υπάρχει μια αυξανόμενη διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να πάρει την πρωτοβουλία για νομοθετικές διαδικασίες όπου η Κομισιόν δεν βλέπει να υπάρχει κάποια ελπίδα να εξασφαλίσει την έγκριση του Συμβουλίου. Η πιο πρόσφατη χρονική περίοδο λοιπόν χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη εφαρμογή και στην διευκρίνηση ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η Κομισιόν έχει την τάση να εστιάζει σε αυτά τα θέματα πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν αλλά μαζί με τους συναδέλφους μου βρήκαμε ότι υπήρξε και σημαντική πρόοδος σε ορισμένα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη για την οδηγία για τα γραφεία προσωρινής εργασίας και για την οδηγία για τα εργασιακά συμβούλια, όπου υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι με την βοήθεια και των κοινωνικών εταίρων. Αλλά γενικά μειώνεται το τμήμα της νομοθεσίας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην διαφάνεια 11 βλέπετε μία σειρά από θέματα τα οποία είναι εκρεμή αυτή τη στιγμή, είναι θέματα τα οποία εξακολουθούν να είναι ανεπίλητα σε μεγάλο βαθμό και παραμένουν επιτάπητος. Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεως στο νομοθετικό πλαίσιο με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπω η οδηγία για το χρόνο εργασία παραμένει ακόμα εκκρεμή η έγκρισή τη. Υπήρξαν κάποιε εξέλιξει σε σχέση με την οδηγία για τι συλλογικέ απολύσει και την μεταφορά επιχειρήσεων, για την ε, ε, μεταβιβασιμότητα των συντάξεων, το θέμα της διευκρίνησης οδηγίας ε, για τους αποσπασμένους εργαζομένους, το οποίο παραμένει στην ημερήσια διάταξη μετά από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επιβάση της παλιάς οδηγίας. Έχουμε το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών σε περίπτωση διαμεθοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η ασφάλεια και η υγεία των εγγύων. Υπήρξε η τροποποίηση της οδηγίας για τη γονική άδεια που ενεκρίθησε στις 8 Μαρτίου από το Συμβούλιο. Υπάρχει οδηγία για την συμμεταχείριση και μια σειρά από θέματα που έχει προωθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της ανανεωμένης κοινωνικής ατσέντας από το 2008 επέκεινα σε ό,τι αφορά ελάχιστα πρότυπα προστασίας, προστασία εισοδήματο, νέες μορφές απασχόλησης, ατομικές απολύσεις, κλπ. κλπ. Τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί όλα αυτά τα θέματα μέχρι στιγμής. Τώρα, κάναμε κάποιες συνεντεύξεις και είδαμε το... κάναμε κάποια έρευνα για το ρόλο του Κοινοβουλίου που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Φυσικά τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του Κοινοβουλίου έχει γίνει πιο σημαντικός ε, και πιο ισχυρός. Την τελευταία δεκαετία είχαμε αυτές τις αλλαγές και λόγω των συνθήκων Φυσικά, ο ρόλος του Κοινοβουλίου παίζει ανάλογα με την πολιτική, ανάλογα με τα μέσα και τα εργαλεία. Αν ε, διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στα ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και στην ε, ε, νομοθετική διαδικασία, ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν είναι ο ίδιος, αλλά έχει γίνει πολύ πιο σημαντικό στην τελευταία δεκαετία. Στην απόφαση και η συνήθις νομοθετική διαδικασία, αυτά είναι μεγάλα, ισχυρά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αυτό το Κοινοβούλιο εξαρτάται και από τη θέληση της Κομισιόν να προωθήσει και να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ε, και μερικές φορές είναι δύσκολο να πείσει στην Κομισιόν ε, αν η ίδια δεν θέλει να υποστηρίξει κάποια θέματα. Κάποια διακυβεύματα. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σημαντικό και είχε μεγάλη επιρροή κάθε φορά που υποστηρίζεται από αρκετές κυβερνήσεις και από κοινωνικούς εταίρους. Ε, μία περίπτωση είναι η, υπηρεσία, η οδηγία για τις υπηρεσίες, όπου ενεπλάκει τα μάλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επηρέασε θετικά την τελική εκδοχή της οδηγίας που υιοθετήθηκε. Ε, ο κοινωνικός διάλογος και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού έχει μερικές, ε, μερικούς τομείς ε, όπου το κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται πολύ. Βεβαίως, ε, το κοινοβούλιο μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του και στα νομοθετικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο να αποκαταστήσει κάποιες συμμαχίες με κάποιους φορείς, όχι μόνο στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών, αλλά και εκτός Κοινοβουλίου ε, με το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις, την Κομισιόν και τους κοινωνικούς εταίρους και το ευρύτερο κοινό, ε, αν υπάρχουν ε, διαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχει διάλογος με την Κομισιόν και το Συμβούλιο βεβαίως. Όλα αυτά είναι στοιχεία που επηρεάζουν την προετοιμασία της απόφασης και είναι πολύ σημαντικά. Η έκθεση επίσης μιλάει για το ρόλο των, της κοινωνικής ε, στα πλαίσια της ε, ατζέντα της ε, Λισαβόνας. Φυσικά υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των οικονομικών πολιτικών που απορρέουν από την ατζέντα της Λισαβόνας και τους κοινωνικούς στόχους. Αλλά δεν υπάρχει, όπως λέμε εμείς, ουσιαστική αντίφαση μεταξύ των δύο. Υπάρχουν πολλοί τομεί όπου μπορεί να υπάρξει συμβιβασμό μεταξύ των δύο ε, και οι οικονομικέ πολιτικέ δεν είναι κατά ανάγκη επιζήμιε για την κοινωνική διάσταση. Ε, μην ξεχνάμε επίση ότι τα εθνικά κοινωνικά μοντέλα διαφέρουν και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και η ήπια νομοθεσία είναι κατάλληλο εργαλείο για να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη και να κινηθούν ε, να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους στις ε, πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές και τελικά τις οικονομικές πολιτικές. Επομένως, ε, πιστεύουμε ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι μια καλή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την ετερογένεια των εθνικών ε, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και να κινηθούμε προς μια κοινή κατεύθυνση. Τώρα με την κρίση, βέβαια, απειλείται αυτή η διαδικασία φυσικά θα επηρεάσει και την νέα στρατηγική με χρονικό ορίζοντα το 2020 που ξεκινάει φέτος. Φυσικά θα πρέπει να ξαναδούμε κάποια παλιά εργαλεία, να τα βελτιώσουμε, να τα αναθεωρήσουμε, ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική. Εργαζόμαστε επίσης για λογαριασμό αυτής της ε, Επιτροπής, αναλύοντας τη σταθερότητα των ε, κοινωνικών πολιτικών μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης. Προσπαθούμε να δούμε όχι μόνο το κόστος, αλλά και το όφελος των κοινωνικών πολιτικών, ε, όπου στα πλαίσια της κρίσης η ανεργία πολύ πιθανόν να αυξηθεί. Υπάρχει και μια νέα απειλή αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας και της αδράνειας στα νέα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με κάποιες ιδέες, με, κάποιους, με κάποιες προτάσεις, όπου νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτές τις ιδέες. Καταρχάς, οι εσωτερικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επιτυχές στις προσπάθειές του όταν είναι συνεκτικό όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων. Ένα άλλο μοχλός επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι αρμοδιότητες για τον προπολογισμό. Οι δημοσιονομικέ αποφάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθούν και να προωθηθούν οι στόχοι τη κοινωνική πολιτική. Επίση, ο συντονισμό με άλλου ε, εταίρου και φορεί είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμπλακεί περισσότερο και πιο ουσιαστικά στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού σε, από την αρχική, από την πρώτη φάση, ε, αποκαθιστώντας ένα μόνιμο διάλογο με την ε, Επιτροπή για να αναπτύξει και να προωθήσει από την πρώτη φάση, από την αρχική φάση της απόψης του για την κοινωνική πολιτική. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα τώρα να σπρώξει την ε, Ένωση να ξεκινήσει διαδικασίες, νέες διαδικασίες νομοθετικές. Και να θέσει κάποια θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο που το απασχολούν. Μπορεί επίσης να ασκήσει περισσότερη επιρροή λόγω των αυξημένων δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων του. Επίσης, κάτι που ήδη είπαμε, να δημιουργεί συμμαχίας με άλλου φορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Συμβούλιο, άτυπο ή επίσημο διάλογο με τα κράτη-μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια, με τους κοινωνικούς εταίρους και τέλος και σημαντικό, ε, την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. τον τρόπο μπορεί να προωθήσει τα θέματα του και αυτοί να το βοηθήσουν. Όλοι αυτοί οι φορεί να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο να τα προωθήσει. Αν δηλαδή ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη, είναι πολύ πιο εύκολο για το Κοινοβούλιο να προωθήσει τα θέματα του. Τώρα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κινείται γύρω από θέματα που είναι ακόμα εκκρεμή. Κάποια είναι ήδη στην ατζέντα, σε κάποια θα σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος από κάποια άλλα. Οι πιο στενές ε, σχέσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν που σας είπα ήδη είναι πολύ σημαντικές και απαραίτητες για να ξεπεραστούν τα διέξοδα. Η σημερινή Ισπανική Προεδρία θέλει να κλείσει την ε, τρέχουσα κοινωνική ατζέντα. Κάποια θέματα λοιπόν φέτος είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και θα υπάρξει μια νέα κοινωνική ατζέντα στο μέλλον. Κάποια θέματα λοιπόν θα τα ξαναδούμε, θα επανεμφανιστούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει σε πρωταρχική ε, φάση να τα επηρεάσει. Τώρα πιο γενικά για τους προσανατολισμούς υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστούν οι ρόλοι των αρχών της ε, αγοράς ε, σε αντιδιαστολή με τα κοινωνικά θέματα και να επιληθούν ε, κάποιες από τις εγγενείς εντάσεις ε, αγορά και ανάπτυξη αγοράς από τη μία και μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές πολιτικές αλλά και εθνικές ασφαλιστικές δικλείδες για κάποιους τομείς όπου οι δημόσιες υπηρεσίες ε, και τα δημόσια Έχω θέσει μάλλον κάποιες ε, οδηγίες εδώ, η οδηγία για τις υπηρεσίες, ε, η απόσπαση των εργαζομένων, οι κοινοφιλείς υπηρεσίες, οι, κοινο... οι πολιτικές ε, αγοράς, εργασίας και κοινωνικές πολιτικές δεν έρχονται σε αντίφαση με τις οικονομικές πολιτικές. Θα εξασφα... Ο συνδυασμός μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική συνοχή και να μην έρχεται σε αντίφαση, αν, όχι να... αν δεν μπορεί να υποστηρίξει τον οικονομικό δυναμισμό. Μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά θα είναι σημαντική για να υπάρχουν ε, ελάχιστα πρότυπα και για να υπάρχουν εθνικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υποσκαφθούν ε, τα κοινωνικά θέματα που είναι σημαντικά και θεμητό να προστατευτούν. Συμπεράσματα. Ε, έχουμε τον ορίζοντα του 2020 μπροστά μας. Αυτή η νέα στρατηγική για το 2020 ε, κινείται προς την κατεύθυνση της ε, ατζέντα της Λισαβόνας. Ε, απασχόληση, πλήρης απασχόληση, ε, δεξιότητες, βίωση της φτώχειας. Αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι ε, τα οικονομικά μελήματα είναι τα κυρίαρχα. Η διακυβέρνηση είναι κάτι που απασχολεί πολύ τη στρατηγική. Ε, για να υπάρξουν και αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο για του συμπεφωνημένου Ευρωπαϊκού στόχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ζητήσει συνεκτικέ πολιτικέ. ίδια προτεραιότητα στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τα θέματα των εθνικών δεσμεύσεων και κατά πόσο είναι αξιόπιστες αυτές. Οι κοινωνικές πολιτικές δεν έρχονται σε αντίφαση κατά ανάγκη με τις οικονομικές πολιτικές υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε στο μέλλον πιο βιώσιμες κοινωνικές πολιτικές, εκπαίδευση, περίθαψη των παιδιών, έβελξη ασφάλεια, κινητικότητα και δυνατότητα απασχόληση του πληθυσμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να επηρεάσει και να παρακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μεταρρύθμισης σε από, την, από τα πρώτα τη βήματα. Αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξει και μεγαλύτερο ρόλο στα πλαίσια του, της μεθόδου συντονισμού. Θα πρέπει να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερη εμπλοκή σε τομείς που δεν διέπονται από την ε, νομοθεσία, αλλά από τη λεγόμενη ήπια νομοθεσία. Επίση, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνδέσει τα κριτήρια κοινωνική πολιτική με τι ε, δημοσιονομικέ αποφάσει. και να προωθήσει πραγματικά τα θέματά του. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, στα πλαίσια της ε, σημερινής κρίσης, μπορεί να, δώσει, μπορεί να προσδώσει μια νέα νομιμότητα στις κοινωνικές πολιτικές. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ουσιαστική πρόοδο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ πριν να δώσω το λόγο στους, ε, ε, στα μέλη, ε, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιο ε, χρονοδιάγραμμα σχετικά με το θέμα του συντονισμού. Ε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μας πείτε ε, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτός ο τομέας. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρξει συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είχε εξαγγελθεί εξ αρχής. Θα ήθελα να δούμε γιατί δεν υπήρξε ε, κάποια, κάποιο επίτευγμα σε αυτή τη φάση και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Επίσης είπατε ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο συντονισμό συντονισμός μεταξύ ε, διαφόρων επιτροπών και ε, μέσα στο Κοινοβούλιο. Εγώ περιμένω πολλά από αυτά. Ίσως θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε, ανάλογα με την θέση που παίρνετε εσείς, πού τοποθετούνται τα προβλήματα, εάν ταυτίζετε την έλλειψη της συνεργασίας ορισμένων, μεταξύ ορισμένων επιτροπών, ή αν νομίζετε ότι ορισμένες επιτροπές συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Ε, ίσως ε, θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Μανπότα και στη συνέχεια θα πάρω όλους τους ε, εγγεγραμμένους αγορητές στον κατάλογο και μετά θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έκθεση. Στην σελίδα 13 αναφέρονται όλα αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για μια περαιτέρω συνεργασία. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας ασχολείται με τα θέματα κοινωνικά και τα θέματα απασχόλησης και έχει προσπαθήσει να προχωρήσει προς συμβιβαστικές λύσεις και νομίζω <clears throat> ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμες όλες οι προσπάθειες που μας δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς και να αποκομίσουμε καλά αποτελέσματα. Χθες είδαμε ότι μπορούμε πάντα να προχωρούμε προς την κατεύθυνση των συμβιβασμών. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται, είναι πολύ σημαντική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες ομάδες που εμπλέκονται στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Είναι σημαντικό για μας λοιπόν να αλλάξουμε μία σειρά από διατάξεις οι οποίες βρίσκονται στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων ήταν θετικό, παραδείγματος το, οποίο, το ότι γεγονός ότι εμείς θεσπίσαμε ορισμένες αρχές για την παροχή υπηρεσιών, ότι εγκρίναμε οδηγίες όπως αυτές για το REACH στο παρελθόν. Και επομένως νομίζω ότι στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής έχει επιτύχει πάρα πολλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτά βέβαια χωρίς χρηματοδότηση, αυτό είναι γεγονό. Πολλές φορές νομίζει κανείς ότι η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού είναι μια τελείως χωριστή υπόθεση και η κάθε Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για τα χρήματα. Αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς δεν είμαστε ένα ταμείο. Εμείς έχουμε την κύρια ευθύνη για θέματα όπως αυτά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε και την επιτυχία των μικρο πιστώσεων. Είναι σημαντικό να υπάρξει και συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτή την πρωτοβουλία. Το Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων φτάνει, έχει μια συμμετοχή στις μικροπιστώσεις ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να γίνουν συγκεκριμένα εγχείρηματα. Έχω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο αφορά ορισμένες βασικές αρχές. Υπάρχει η Ατζέντα 2020 από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φαίνεται σαν μια φρικτή γραφειοκρατική ρύθμιση. Εμείς όμως θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε και κάποιες βασικές ιδέες, έχουμε ένα όραμα με το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε τη στρατηγική του 2020 σε μια καθαρά γραφειοκρατική αντιμετώπιση, ένα γραφειοκρατικό εγχείρημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να τη συνοδεύεται αυτό από ένα σύνθημα, από ένα όραμα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Τέλος, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα της κατάρτισης, όπου δεν έχουμε καταφέρει να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Παραγωγή χάρη σε ό,τι αφορά τα οικολογικά θέματα, είναι απαραίτητο να μπορέσει να υπάρξει μια αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων. Είναι το πιο δύσκολο αυτό, να μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη, να του πούμε ότι πράγματι πρέπει να προχωρήσετε σε αυτόν τον τομέα. Θέλουμε να διατηρήσουμε μεν την επικουρικότητα, βεβαίω, Θέλουμε όμω να έχουμε και περισσότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ μα. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου, πιστεύω. Γιατί είναι πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία κρατούν μια στάση αμυντική, μια στάση κατανάτσιο. Εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών να μπορέσουμε να μάθουμε αμοιβαία ημένα από τους δε, να αναπτύξουμε περισσότερη ανταλλαγή απόψεων και μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-μέλη και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πάντα έτοιμοι να μάθουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κινητοποιήσουμε τους άλλους. Λοιπόν, θεωρώ ότι η μελέτη αυτή ήταν μια πολύ καλή ανάλυση. Ευχαριστώ κύριε Θέρκας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στον προβληματισμό που έκανε ο κύριος Μαν. Μου, είναι, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβούμε σε αυτή την προβληματική, στον προβληματισμό, αλλά θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της έκθεσης που εγώ την διάβασα πολύ προσεκτικά. Είναι πολύ θετικό κάποιο, έξω από εμά που είμαστε οι νομοθέτε, να μπορέσει να αξιολογήσει και να αποτιμήσει αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και να μα δώσει κάποιε κατευθύνσει σκέψει να μα πει πού είναι τα ισχυρά και πού είναι τα αδύνατα σημεία τη δράση μα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την κοινωνική ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι μονάχα θέμα πολιτικών, αλλά είναι και απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι αυτές οι πολιτικές βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης για να μπορέσει να υπάρξει και ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιφαλλοντικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμμετέχω λοιπόν και αποδέχομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν σε αυτή την ε, έκθεση και συμμερίζομαι και αυτά που είπε ο κύριος Μάν για την στρατηγική του 2020. Θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική η οποία δεν παραγνωρίζει την κοινωνική διάσταση και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή την πορεία. Θα ήθελα απλώς να πω ότι από μια ε, επιπόλαια κάπως ανάγνωση αυτού του εγγράφου πιστεύω ότι ακόμα χρειαζόμαστε, δεν ξέρω αν αυτό είναι το δικό σας καθήκον ή κάποιον άλλον, χρειάζεται να έχουμε ένα καλύτερο όραμα και μια καλύτερη αποτίμηση της πολιτικής κοινωνικών θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο να σε ό,τι αφορά το ρόλο που έχουν παίξει τα θεσμικά όργανα και οι άλλοι παίκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την έποψη του ποια είναι τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε σε αυτό το μικρό κόσμο των Βρυξελών, το Συμβούλιο Κομισιών και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υπάρχει λοιπόν μια επιτό, μια αποτίμηση καλύτερα του πώς αντιμετωπίζει ο απλός άνθρωπος τους παίκτες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Είπατε ότι είναι απαραίτητη μια πολιτική συμμαχιών για να μπορέσουν να προωθηθούν αυτά τα οποία θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφερθήκατε σε μια πολιτική συμμαχιών με την κοινωνία των πολιτών. Θα μπορούσατε κάποια στιγμή να αξιολογήσετε, υπάρχει κάποιο τρόπο να αξιολογήσουμε το πώ βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτε την πολιτική που ασκείται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο όχι σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μοντέλο που ξέρουμε ότι είναι αρκετά ετερογενείς οι εθνικές πολιτικές, αλλά να καταλάβουμε πώς βλέπουν οι πολίτες σε αυτό το θέμα, την ευρωπαϊκή διάσταση στα κοινωνικά θέματα, την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης. Όχι μόνο λοιπόν να μιλάμε για προβλήματα, αλλά να μπορέσουμε να διακρίνουμε πού βρίσκονται τα συμβούλια. Παραδείγματο χάρη, για την οδηγία χρόνου εργασία Μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Εμά μας φάνηκε ότι αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στο επίπεδο τη νομοθετική ε, οικοδόμησης της Ευρώπης. Αλλά μπορεί τελικά στην κοινή γνώμη να φάνηκε ότι ήταν λαθασμένη αυτή η νομοθεσία. Καλύτερα να υπάρχει νομοθετικό κενό για μένα παρά νομοθεσία η οποία θα είναι λαθασμένη και όχι αποδεκτή από την κοινωνία. Είναι λοιπόν η στιγμή να υπάρχει ένα καλύτερο διάλογο και είναι η στιγμή να καταλάβουμε ότι ο κόσμο των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο πραγματικό κόσμο. Ο πραγματικό κόσμο είναι αυτό ο οποίο βρίσκεται έξω από τα τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα πως το δικό μας έργο επηρεάζει την καθημερινή πραγματικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων γιατί φοβάμαι μερικέ φορέ ότι έχουμε μια μεγάλη αυτοικανοποίηση με το έργο το οποίο κάνουμε εμείς, αλλά κάθε πέντε χρόνια μας λένε ότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάνετε και κανείς δεν καταλαβαίνει τι κάνετε. Μας βλέπουν οι πολίτε σαν απομακρυσμένου από την πραγματικότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να σα ευχαριστήσω για την πάρα πολύ σημαντική αξιολόγηση που κάνατε που αναφέρεται τα θετικά και τα αρνητικά σημεία τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα πραγματικά όμω να έχω και περισσότερα στοιχεία. Θα έκανε τέλειο το έγγραφο αυτό αν μα λέγατε πώ μα βλέπουν όχι μονάχα οι εμπειρογνώμονε και οι ερευνητέ, αλλά και ο απλό πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν, πρωτού επανέλθω στου ομιλητέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον συγγητή αυτής της έκθεσης. Ε, ε, διάβασα μόνο τις δύο-τρεις πρώτες σελίδες ενδελεχώς, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κείμενο, φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο για την εργασία μας. Θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Μόλις επικυρώσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και ένα από τα θέματα που θίγεται στην εισήγησή σας είναι το πώς παρακολύονται οι υποθέσεις στο Συμβούλιο. Ε, υπάρχει το θέμα της ψηφοφορίας με πλειοψηφία και το πώς αντικατοπτρίζεται η επίπτωση αυτού του προβλήματος στις διάφορες υποθέσεις που διεκπεραιώνονται. Θα υπάρξει βελτίωση όταν υπάρξει βελτίωση και της νομοθεσίας. Θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να ακούσω μια απάντηση σε αυτό το σημείο. Επίσης, μιλάτε για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για το πώς ε, ε, πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό να είναι υποχρεωδεσμευτική η θέση του Κοινοβουλίου στη συμμετοχή του και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν το εξετάσαμε ικανά μέχρι στιγμής. Έχετε κάποιες προτάσεις ενδεχομένως για το πώς θα καταρτιστεί όλος αυτός ο μηχανισμός για να υπάρξει ένα σωστό ε, πλαίσιο καθοδήγησης και τι θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να, να πράξει όταν θα του ζητηθεί να συμμετάσχει ε, σε αυτή τη διαδικασία διαδικασία και ύστερα πηγαίνοντας ε, στην, στον στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού λέτε ότι πρέπει να βρεθούν ελάχιστες προδιαγραφές για την, το, τις κοινωνικές υπηρεσίες στο κράτος πρόνοιας, στο κράτος εμπάρειας κτλ. Και λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει ε, δυσχερέστερες τις διαδικασίες. Ίσως θα πρέπει να το εξηγήσετε αυτό. Πώς το βλέπετε, κατανοώ τι εννοείτε, αλλά θα ήθελα να ε, μας φωτίσετε λίγο περισσότερο. Επίσης, Επίσης ε, ε, λέτε ότι ενώ χρειαζόμαστε ε, αξιολόγηση του, της πολιτικής ατζέντα, πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει αυτή και πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να διευκρινιστεί. Επίσης ε, το θέμα είναι η κοινωνική πολιτική της ΕΕ. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ε, ίσως να, ξεκινήσουμε πολύ να ξεκινήσαμε πολύ ισχυρά στην δεκαετία του 70 και του 80 με το Βερολίνο που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά αλλά υπήρξε μια επιβράδυνση ως προς το κοινωνικό μοντέλο. Και θέλω να ξέρω και εδώ τη γνώμη σας. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω και να σας ρωτήσω για το ποια είναι η γνώμη σας είναι πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσουν ορισμένες υποθέσεις. Έχετε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες πάνω σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις αρμοδιότητες και την εξουσία μας σε αυτό το τομέα, ούτω ώστε να έχουμε μια διαφορετική θέση. Έχετε κάποια ιδέα τι θα μπορούσαμε, πώς θα μπορούσαμε να συμπράξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκοστά, ευχαριστώ για τα πολύ βοηθητικά σας σχόλια. Ε, ο, ορισμένα έχουν ήδη καλυφθεί ε, ε, στα, ως προς τα διάφορα θέματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ ή όσο καλύτερα μπορούμε αν θέλετε θα παρουσιάσουμε ε, μια στήριξη των διαφόρων πολιτικών που έχουν σχέση με την κρίση. Ε, επίσης το θέμα του ε, κόστους και της επεξεργασίας του ρόλου που έχει εγκριθεί για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και την χρηματοοικονομική πολιτική και πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι τύποι ε, εργαζομένων οι οποίοι καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση αλλά ε, ωστόσο υπάρχουν οι προσωρινοί εργαζόμενοι, οι ε, μερικώς απασχολούμενοι κτλ οι οποίοι δεν καλύπτονται και είναι δύο κατηγορίες ε, εντελώς διαφορετικές και επίσης το θέμα του ΠΟΕ ε, είναι ένα θέμα που ανήκει στον πυρήνα της όλης διαδικασίας είναι κάτι το οποίο το έχετε θέσει και εσείς κυρία Πρόεδρε και ο Ιρλανδός συνάδελφος και νομίζω ότι βασικά έχουμε ορισμένες πολύ ε, θετικές γνωστές απόψεις. Το Κοινοβούλιο δέχεται ε, ε, διάφορες νομοθετικές συμβουλές πριν να εκπονήσει τις νομοδοτήσεις του και προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις καταστάσεις σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη της Κομισιόν, δηλαδή τι θέματα βάζει στην ημερήσια διάταξη η Κομισιόν όταν καταρτίζεται η επίσημη ημερήσια διάταξη που θεσπίζει το διάλογο ανάμεσα στην Κομισιόν και τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα πυρηνικού χαρακτήρα. Επίσης ε, υπάρχουν ορισμένες νομοθεσίες οι οποίες ε, δεν έχουν πλήρως ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Θα αυτό πρέπει να γίνει στο μέλλον. Τώρα για τη συνεργασία των διαφόρων επιτροπών μεταξύ τους, εδώ βλέπετε ότι έχετε εσείς περισσότερη συνέστηση των προβλημάτων από μένα. Ενδεχομένως θα πρέπει να πούμε ότι ε, υπάρχει μια ρήτρα συντονισμού η οποία θα μας ωφελήσει ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία στο Κοινοβούλιο για την εκπόνηση ορισμένων θέσεων, για την εσωτερική αγορά για παράδειγμα. Υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές που αφορούν και τους κανονισμούς ε, που διέπουν την ε, εσωτερική αγορά. Φαίνεται να είναι αρχικά απομονωμένα αυτά τα πεδία, αλλά υπάρχουν ευρύτερες οικονομικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότερο ή λιγότερο εξάλλου πάνω ε, στο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε από κοινού ε, και πώς μπορούμε να βρούμε συμβιβασμούς ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στους άλλου θεσμούς. Είχαμε interviews με τους παρατηρητές, συζητήσαμε μαζί τους και είδαμε ότι όλοι συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση ότι είναι καλύτερα να υπάρχει νομικό κενό από το να υπάρχει νομοθεσία που δεν είναι ικανοποιητική για τους πολίτες, κακή νομοθεσία. Και επίσης υπάρχει κάποιο κόστος για την εκπόνηση της νομοθεσίας με οποιοδήποτε τίμημα. Ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει θέση πάνω σε αυτό, να έχει μια όσο πιο ισχυρή και καλή θέση και επίσης να υπάρχει κάποιος ρεαλισμός για ορισμένα θέματα τα οποία θεωρούμε με θέματα προτεραιότητας και όπου χρειάζεται να γίνουν ορισμένοι ε, συμβιβασμοί για το τι πρέπει να επιτευχθεί, τι πρέπει να γίνει. Και ο συνάδελφός μου, ο Μάικολ, ίσως θα ήθελε να πάρει το λόγο ε, από αυτού. Ευχαριστώ κύριε Μαν. Η Ευρώπη 2020, δηλαδή του 2020, θα ασχοληθεί με την οικονομία και την αύξηση, οικονομική στρατηγική και στρατηγική αύξηση. Ε, έχουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις ε, πάνω σε κοινωνικά θέματα όπως είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και ε, η μείωση της ενέργειας και εάν δούμε αυτόν τον τομέα πρέπει να γίνει πιο σωστός καθορισμός των κοινωνικών θεμάτων πιστεύω, πιο επακριβή σε ό,τι αφορά τη σχετική στρατηγική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Ε, θέλετε να υποβάλλετε κάποιο άλλο σχόλιο πριν να δώσω το λόγο σε άλλους ομιλητές. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι ε, για τον κύριο Σέρκα πρέπει να πω ότι ευχαριστώ για τα σχόλια του και χαίρομαι όταν το Κοινοβούλιο προτείνει μια ισότιμη εξέταση των ε, κοινωνικών στόχων και σε θέματα νομοθεσίας αλλά και σε θέματα εφαρμογής και βεβαίως ε, όλα όσα καλύπτουν την εξωτερική αντίληψη του τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια είναι τα επιτεύγματα, ποιε είναι οι δράσεις τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτά θα ζητήσουν θα απαιτήσουν μία άλλη επισκόπηση της στάσης των πολιτών αν θέλετε ε, ως προς την Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά κάποιο τρόπο να δούμε πώς αντικατοπτρίζονται οι απόψεις μας, σε ποιο βαθμό το έργο των ε, θεσμικών οργάνων αναγνωρίζεται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Ε, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα από αυτά τα θέματα για τις ελάχιστες προδιαγραφές. Νομίζω ότι αυτό το θέμα ε, για να το δούμε θα πρέπει να ε, εξακριβώσουμε ότι υπάρχει ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θεσμικά όργανα και οι οικονομικές επιδόσεις είναι πολύ ποικιλόμορφες και αυτές είναι άνισες για τις ελάχιστες, για τις ελάχιστες προϋποθέσεις ε, θα πρέπει να υπάρχει μία λύση σε σχέση με αυτές ούτως ώστε να αποφύγουμε ορισμένες υπερβολικές επεκτάσεις της αγοράς με ανερχό τρόπο. Θα μπορούσε να είναι αυτή μια ρεαλιστική, πραγματιστική προσέγγιση, να υπάρχει μια ομοιογένεια και όχι ετερογένεια ε, σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα. Ορισμένα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να μπουν σε μια ημερήσια διάταξη που να ασχολείται με θέματα που αυτή τη κατεύθυνση. αυτή της κατεύθυνσης. Δηλαδή να υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας, να αποφασιστεί αυτό το επίπεδο προστασίας και ε, να μπορούμε εμείς να εισαχθούμε σε ένα πλαίσιο με έναν κοινό τρόπο ε, με τα κράτη-μέλη ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων πόλων ε, μέσα στην κοινότητα και να εκμεταλλευτούμε τα θετικά, τον ανταγωνισμό θετικά των κρατών μελών μεταξύ τους. Όπως ξέρουμε υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια θεσμική συμφωνία μεταξύ των δύο οργάνων ε, για το δικαίωμα το απεριόριστο να υπάρχουν αιτήματα για νομοθετικές προτάσεις σε κάτι το οποίο το επιβάλλει η Επιτροπή και αυτό έχει ε, αυξήσει το κόστος της ε, ε, Επιτροπής σε ό,τι αφορά την απόρριψη των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και προτείνει νέες υποθέσεις. Και ίσως θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δυνητικού κινητήριου μοχλού της ατζέντα για τα κοινωνικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι εσείς πράγματι έχετε αρκετή επιρροή για να μπορέσετε να φέρετε στο προσκήνιο ορισμένα από τα θέματα τα οποία θεωρείτε εσείς σημαντικά και χρήσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια σχόλια λοιπόν σχετικά. Θα πρέπει να γνωρίζει κανείς και τους περιορισμούς της δημιουργίας ε, συμβιβασμών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένες φορές μπορεί να είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι λυσιτελές, να εστιάζει κανείς την προσοχή του μονάχα σε ορισμένα εφικτά ζητήματα για να μην υπάρξει η αρνητική στάση της Κομισιόν ή του Συμβουλίου. Θα πρέπει κανείς τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για να μπορέσει κανείς να προωθήσει μια σωστή νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τουρόν, κυρία Μοράλ, ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Δανέζικα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη στην οποία προχωρήσετε. Δεν την έχω διαβάσει ενδελεχώς. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα τα οποία ε, εμένα μου έχουν δημιουργήσει προβλήματα ως νέο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σε επίπεδο προσόντων και ένα μεγάλο χάσμα σε ό,τι αφορά τα θέματα εσωτερικής αγοράς από τη μια μεριά και των κοινωνικών θεμάτων. Εγώ ανήκω στην Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς όπου τονίζουμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια κοινή πορεία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οικονομικό τομέα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσει κανείς όλα αυτά τα μέτρα, τα νομοθετήματα και υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία έλλειψη που οφείλονται στο γεγονό ότι δεν υπάρχει απόλυτο συντονισμό της ε, κοινωνικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής με την πολιτική ε, οικονομικών θεμάτων. Υπάρχει και ένα χάσμα επίσης σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, γιατί η Κομισιόν έχει ένα πολύ έντονο κάθετο χαρακτήρα μέσα στις αρμοδιότητές της και είναι ίσως σε στεγανά οργανωμένες οι υπηρεσίες της. Θα ήθελα να, λοιπόν να σκεφτώ, να, να, να ακούσω την άποψή σας πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το χάσμα, να έχουμε λιγότερα στεγανά και για το αν θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα πρωτοβουλία σε επίπεδο ήπια νομοθεσία. Σε όλη τη στρατηγική του 2020 το Κοινοβούλιο είναι παραμερισμένο ουσιαστικά. Εγκρίναμε στο Στρασβούργο ένα ψήφισμα το οποίο ήταν πολύ νερωμένο και αποδυναμωμένο για να έχουμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων τελικά αυτό το οποίο βγήκε είναι τόσο αδύνατο και ισχνό που ουσιαστικά δεν λέει τίποτα στην Κομισιόν. Δεν λέει τίποτα το οποίο δεν ξέρει. Είναι απαραίτητο όπως λέτε να σφυριλατήσουμε συμμαχίες. Ωραία. Αλλά είναι αυτό αρκετό για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά επιρροή στις μεγάλες στρατηγικές οι οποίες θα αναπτυχθούν τα επόμενα δέκα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει διαδραματίσει το ρόλο τον οποίο έχει, έπρεπε να αναφέρει και επίσης ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για τον προϋπολογισμό. Uh, ευχαριστώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συντάκτες ε, της μελέτης ε, γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε μία αναδρομή στο πώς ε, δουλέψαμε, τι καταφέραμε για τη στρατηγική της Λισαβόνα στην περίοδο 2000-2010. Όλοι γνωρίζουμε ότι για να επιτύχει η κοινωνική ατζέντα υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δουλέψει κανείς ο δικός μας, από τη μία, αλλά από την άλλη η εξωτερική επίπτωση της κρίσης ε, παρεμπόδισε την υλοποίηση των στόχων που είχαμε θέση. Αυτό αποδεικνύει ότι τα οικονομικά ζητήματα, είτε μας αρέσει είτε, δεν μας αρέσει, έχουν σοβαρότατη επίδραση πάνω στις κοινωνικές πολιτικές. Για τη στρατηγική του 2020, λοιπόν, όσο δεν έχουμε απορροφήσει την κρίση και εξέλθει από αυτήν, οι κοινωνικές μας ε, πολιτικές θα είναι ευάλωτες και οι στόχοι θα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Συνολικά τώρα, για τον τρόπο εργασίας, για τον τρόπο που δουλέψαμε, είπαμε πάρα πολλά. Είπαμε πολλά για την ε, άποψη των, και την αντίληψη των ε, πολιτών. Ίσως δεν υπάρχει αυτό το θέμα στη μελέτη σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτή τη στάση. Πρέπει μέσα από τις κοινωνικές πολιτικές που πραγματικά επηρεάζουν τους πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, μέσα από αυτές οι συμπολίτε μας θα, θα αντιληφθούν την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει η Ευρώπη μέσα από τα θεσμικά όργανα που δεν τους ενδιαφέρουν και τόσο, παρά μέσα από τις κοινωνικές πολιτικές και τα ωφέλη τους. Δεν πρόκειται για μελέτη για τις απόψεις και τις τάσεις, όπως είπατε, απαντώντας τον Αλεχάνδρο Σέρκας. Το θέμα είναι πώς θα γνωρίσουμε την Ευρώπη στους συμπολίτε μας μέσα από την κοινωνική πολιτική. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να αντιδράσετε σε αυτό που είπα. Δεύτερον, Μας έδωσε συμβούλιο, ε, μια συμβουλή. Ε, μας προτείνεται να συνεργαστούμε τα θεσμικά όργανα μεταξύ μας και να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη ε, και κυρίως με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Μετά από αυτά που είπε η Έμιλη Τουρουνέν, θα ήθελα να θέσω κάτι άλλο, το οποίο δεν θίξατε. Μήπως θα πρέπει να συνεργαστούμε και με ένα άλλο επίπεδο στο εσωτερικό των κρατών μελών, που είναι πολύ σημαντικό για τις πολιτικές μας, το περιφερειακό επίπεδο. Φυσικά πρέπει να έχουμε άμεση επαφή με το εθνικό επίπεδο για να καθορίσουμε τους μεγάλους προσανατολισμούς και για να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο οι πολιτικές μας. Αλλά αν θέλουμε να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών, νομίζω ότι το κατάλληλο επίπεδο είναι το περιφερειακό. Δεν είπατε τίποτα για το θέμα αυτό. της συνεργασίας και της επαφής που πρέπει να έχουμε με το περιφερειακό επίπεδο. Αλλά νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Σας θέσω λοιπόν αυτό το ερώτημα. Θα πρέπει να είμαστε στον πιο κοντά στο επίπεδο που εφαρμόζονται οι πολιτικές μας. Και νομίζω ότι είναι και μια απάντηση για να υπάρξει μια ανάσχεση της απομάκρυσης της Ευρώπης από τους πολίτες. Έπειτα, το τρίτο θέμα συνδέεται με αυτό που είπε ο Τόμας Μαν. Ότι δεν εναρμονίσαμε το περιεχόμενο των διπλωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ό,τι και να πούμε για τη στρατηγική 2020, για την κινητικότητα των νέων, για την πλήρη απασχόληση, για το ευρωπαϊκό χώρο ζωής και εργασίας, ό,τι και να πούμε, αν δεν συμφωνήσουμε πολύ γρήγορα τα 27 κράτη-μέλη επί του ορισμού του περιεχομένου των διπλωμάτων, κάτι που συνδέεται με τον προσδιορισμό των επαγγελμάτων, δεν νομίζω ότι πρέπει να επιτύχουν οι κοινωνικές πολιτικές ευρωπαϊκής κινητικότητας κινητικότητας, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, τι στρατηγικές θα υλοποιήσουμε. Αν ε, συμφωνούμε επί του πολιτικού στόχου, πρέπει να δούμε τι στρατηγικές θα εφαρμόσουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα οι νέοι στην ε, Ευρώπη. Ε, τι αντίληψη έχουν για την Ευρώπη, υπάρχει κινητικότητα, πώς μπορούν να μπουν στον, ε, στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα λοιπόν του περιεχομένου των διπλωμάτων τους, νομίζω τουλάχιστον ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να υλοποιήσουμε αυτό το στρατηγικό στόχο που είναι πραγματικά πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Τσίμερ και κυρία Φιγκερέιδο. Ε, Ευχαριστώ πολύ τους παρουσιαστές. Ευχαριστώ πολύ τους αυτής της μελέτης και φυσικά για την έρευνα που έχουν ε, κάνει για να μπορέσουν να καταλήξουν στο έγγραφο που μας παρουσίασαν σήμερα. Εγώ μπορώ να δώσω μόνο δίκιο στην κυρία Τουρούνεν. Είμαι πέντε χρόνια στο, στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Θέλω να τονίσω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να έχει κανεί μια γενική επισκόπηση για το πώ λειτουργούν αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα εθνικά κράτη. Πού ακριβώ ασκείται η κοινωνική πολιτική είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κανεί. Υπάρχει λοιπόν μια ασάφεια σε σχέση με το πού ακριβώ θα πρέπει να δοθεί η έμφαση αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει τα πράγματα. Από αυτή την άποψη η μελέτη σα είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί ουσιαστικά καταδεικνύει την αλληλεπίδραση σε διάφορα επίπεδα και μεταξύ διαφόρων εργαλείων. Γι' αυτό είμαι πράγματι ευγνώμων σε εσά και νομίζω ότι είναι χρήσιμη αυτή για την εργασία μα. Τρία σημεία τώρα θέλω να θίξω. Καταρχήν σε σχέση με τη στρατηγική του 2020. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να καταλήξουμε σε ένα διευρυμένο ορισμό της ένδειας. ακόμα και μέσα στα πλαίσια της Eurostat, θελήσαμε να κάνουμε πιο σαφές τι σημαίνει του να βρίσκεται κανείς κάτω από τη γραμμή ένδειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όταν πρόκειται όμως για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των ε, ορισμών για να αποφασίσουμε τι αποτελεί ή όχι κοινωνικό αποκλεισμό, τα κράτη-μέλη σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορίζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα κριτήρια και ουσιαστικά τα περιορίζουν σε ένα επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων, πληρωμών, επιδομάτων κτλ. Το βλέπουν με καθαρά οικονομικούς όρους. Το έγγραφο του Μπαρόζο για την στρατηγική του 2020 ανέφερε σε πολλά σημεία το ότι η Κομισιόν ότι είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ατόμων που βρισκόταν κάτω από την γραμμή ένδυας. και τόνιζε ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο γενική οικονομική ανάπτυξη αλλά και βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης των, ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό να έχουμε άτομα τα οποία είναι κάτω από αυτή την γραμμή ένδυας. Ο δείκτης αυτός λοιπόν ο οποίος έχει διατυπωθεί από την πλευρά της Γαλλίας για την καταμέτρηση της ένδυας είναι κάτι το οποίο σας βρίσκει σύμφωνος ή όχι. Και επιπλέον εγώ θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια των εργαλείων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός ότι πρέπει αυτοί οι δείκτες να διατηρηθούν και ενισχυθούν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συμφωνία από την πλευρά των κρατών μελών για την σωστή εφαρμογή αυτής της εργαλειοθήκης και των δικτών. Μόνο αν και τα 27 κράτη-μέλη θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα θα πάνε τα πράγματα καλά. Είναι πολλά τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Επίση, αναφερόσαστε στα θέματα ελαχίστων κανόνων και έχετε εξηγήσει τι σημαίνει αυτό σε εθνικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω όμω ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητε να προχωρήσουμε σε μια στοχοθεσία κριτηρίων. Να καταλήξουμε σε κριτήρια ώστε τα ελάχιστα πρότυπα να ερμηνεύονται μέσα στα πλαίσια των εθνικών συνθήκων. Δηλαδή να περιγράψουμε ένα σύνολο από πρότυπα, από βασικές υπηρεσίες, από κριτήρια, τα οποία τελικά θα είναι εφαρμόσιμα και σε επίπεδο εθνικών κρατών, κάτι το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. όπως παραγωγικά το δικαίωμα για μια βασική πρόσβαση στην ενέργεια. Το θέμα αυτό είχε τεθεί παραγωγικά στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου που είχαν πει ότι θα πρέπει το πολύ το 10% ενός, του εισοδήματο ενό νοικοκυριού να αποδίδεται στην αγορά ενέργειας για να υπάρχει ζεστό νερό, θέρμανση κτλ. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια χρηματοδότηση από το κράτος. Να υπάρξει λοιπόν μια διατύπωση αυτών των βασικών αναγκών και πώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και επίσης το θέμα των εργαλείων που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο να έχουμε και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει κάποια δικαιώματα μέσω κανόνων εφαρμογής, μέσω πολιτικών πρακτικών και σε αυτή την περίπτωση να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου όχι μονάχα στην αντίστοιχη κυβέρνηση, αλλά να υπάρχει και ένα σύστημα προειδοποίησης έγκαιρης το οποίο να εφιστά την προσοχή της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη υπήρξαν άτομα τα οποία πέθαναν από το κρύο στην Πολωνία και στην ε, Γερμανία τον προηγούμενο χειμώνα. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν συστήματα προειδοποίησης ότι ορισμένα άτομα δεν έχουν αρκετή υποστήριξη και υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγικά 100.000 άτομα στη Γερμανία που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το λογαριασμό ενέργειας για να ζεσταθούν. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να περνάνε από τις εθνικές αρχές, από την επικουρικότητα, αλλά θα είναι απαραίτητο οι οποιοδήποτε κανόνες και τα πρότυπα που θα έχουμε να έχουν εφαρμοσιμότητα και να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα και πάλι κάθε χειμώνα όπως στη Ρουμανία, στην Πολωνία και στη Γερμανία έγινε πρόσφατα. Κυρία Φιγκερέιντου. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε τα θέματα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει ήδη και στο παρελθόν, εδώ και πολλά χρόνια. Για μένα εμπεριέχουν ένα πρόβλημα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει καταφανεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές και ιδιαίτερα οι νομισματικές πολιτικές η τάση φιλελευθερωποίησης είτε στην εσωτερική αγορά είτε στα πλαίσια του ΠΟΕ επιβάλλουν πέραν των άλλων πολιτικών και έχουν πάντα τις ίδιες συνέπειες, όπως δείχνει και η πραγματικότητα. Δηλαδή, αύξηση της ανεργίας, αύξηση της ένδυας, όξυνση των ανισοτήτων. Γι' αυτό θέλω να θέσω το εξής ερώτημα η κοινωνική ατζέντα, την οποία εμεί καταφέραμε να έχουμε μέσα στα πλαίσια της δράσης μας, σε τι ωφελεί αν δεν αλλάξουμε το μακροοικονομικό πλαίσιο, σε τι ωφελεί αν δεν αλλάξουμε την νομισματική πολιτική, το σύμφωνο σταθερότητος, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να τηρούν ορισμένου κανόνες, ακόμα και όταν είναι φανερό ότι μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση κρίσης μία περίοδος χαλαρότητος και μετά επανερχόμαστε πάλι στον αυστηρό κορσέ του Συμφώνου Σταθερότητος που οδηγεί σε περικοπές των δημοσίων υπηρεσιών, των αποδοχών των εργαζομένων, επομένως πάλι ένδια και ανεργία. Και το ίδιο αφορά και τις ε, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την κατεύθυνση του ΠΟΕ που οδήγησε στην καταστροφή και στον όλεθρο παραγωγικού τομεί σε πολλές από τις χώρες μας δύο στη δική μου την Πορτογαλία. Αλλά σε ό,τι αφορά και αυτό στην τομέα της γεωργίας και της ε, βιομηχανίας και σε άλλους τομείς. Σας λέω λοιπόν ποια είναι λοιπόν μια κοινωνική ατζέντα που μπορεί να αντέξει σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Λοιπόν αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Ευχαριστώ. Ε, θα ξαναδώσω το λόγο στους ε, ομιλητές του πάνελ. Σχόλια. Ε, Μερικά από αυτά τα θέματα είναι αρκετά περίπλοκα. Αλλά υπάρχουν κάποια light motive που επανέρχονται. Τι σχέση στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, αλλά και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Τη σχέση της ε, εσωτερικής αγοράς με τις κοινωνικές πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές είναι κρίσιμες, όντως και το καλύτερο θα ήταν να κινηθούμε προς μία κατεύθυνση έτσι, μεγαλύτερης ισοτιμίας ε, με τους μηχανισμούς της αγοράς. Οι κοινωνικές πολιτικές δεν είναι μόνο ένα δεκανίκι, είναι ουσιαστικές πολιτικές, είναι βασικές πολιτικές, πυρηνικές πολιτικές οι κοινωνικές πολιτικές και τα κοινωνικά αποτελέσματα είναι προϋπόθεση για την αποδοχή του ευρωπαϊκού στοιχήματος και της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να έχουν αντιρρήσεις εάν ε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση επηρεάζει αρνητικά το βιωτικό τους επίπεδο. Υπάρχει δηλαδή μια αντίληψη της όλης κοινωνίας για την, ε, το ευρωπαϊκό project. Και εκεί εντάσσονται οι κοινωνικές πολιτικές. Φυσικά θα πρέπει να επιτύχουμε μια, τον οικονομικό δυναμισμό και μέσα από αυτές που είναι απαραίτητες σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ε, σε μια τέτοια περίοδο αποκλείεται να ρυθμίσουμε σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο όλε τι κοινωνικέ πολιτικέ. Προφανώ πρέπει να προβλέψουμε κάποια ευελιξία. Πρέπει να την αποδεχτούμε αυτή την ευελιξία. Αλλιώ οι οικονομίε και οι κοινωνίε ε, θα γίνουν φτωχότερε. Φυσικά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ε, παραγωγικές ευκαιρίες που υπάρχουν. Τότε το στίχημα είναι να υπάρξει στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιες αρχικές ασφαλιστικές δικλίδες και να πούμε ότι εκεί οι δυνάμεις της αγοράς δεν πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Παραδείγματος χάρη ελάχιστη μισθή, προστασία του ελάχιστου εισοδήματος, κοινωνικές υπηρεσίες που είναι κρίσιμες και εκ των όνου κάνευ για την αποδοχή του κοινωνικού μας συστήματος. Νομίζω ότι αυτό το είπε και η κυρία Τσίμα στη δήλωσή της. Φυσικά πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσουμε τα ελάχιστα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και μία κοινή συμφωνία σε ευρωπαϊκό, κοινή αντίληψη αν θέλετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι, για το τι παίρνει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης. Τι δικαιούται αν θέλουμε να μειωθεί η φτώχεια μέσω των συστημάτων ε, και προγραμμάτων προστασίας του ελάχιστου εισοδήματο. Ε, χρειαζόμαστε και πολιτικές εκπαίδευση και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρατε την κατάσταση στη Γερμανία για την προστασία του ελάχιστου εισοδήματος. Είπατε ότι ίσως αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Μπορεί. Αλλά κάτι που είναι εποφελές ε, είναι ότι έχουμε το σταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία που μπορεί να πει αυτή η νομοθεσία είναι συμβατή με το Σύνταγμα, η άλλη νομοθεσία δεν είναι συμβατή με το Σύνταγμα. Και πρόσφατα μάλιστα εκδόθηκε μια απόφαση για την καταλληλότητα των προγραμμάτων υποστήριξης του ελάχιστου εισοδήματο. Όχι κατά ανάγκη ότι πρέπει να αυξηθεί το δίχτυ αυτό, αλλά ότι ο υπολογισμός αυτού του ελάχιστου εισοδήματο θα πρέπει να είναι πιο διαφανής, πιο σαφής. Δεν γνωρίζω τη γαλλική συζήτηση για τους δείκτες για τη φτώχεια. Αν μπορούσατε να με ενημερώσετε για το θέμα αυτό, θα ήμουν ευγνώμων για να το συζητήσουμε αργότερα, κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι αυτά αρκούν προς το παρόν. Α, να πω κάτι στην κυρία Τουρούνεν. Είναι σημαντικό να συνδεθούν διάφορες πολιτικές και οι πολιτικές οι οποίες αποφασίζουν για τα οικονομικά θέματα, τα, τον προϋπολογισμό, και τις σκληρές πολιτικές, να, όλες αυτές τις πολιτικές να αφυπνιστούν για τα κοινωνικά θέματα, τα κοινωνικά μελήματα. Και να γίνει μια ε, σοβαρή συζήτηση με την Επιτροπή και τους φορείς που ασχολούνται με την εσωτερική αγορά για τις κοινωνικές πολιτικές. Ο άλλος ομιλητής από το πάνελ θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ εκ μέρους των μελών της ε, Επιτροπής. Θαυμάσια η έκθεσή σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε πότε η ανάλυση κόστους ωφελίας των κοινωνικών πολιτικών θα είναι έτοιμη. Αυτά όμως προς τον παρόν. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στην έκθεση Τσίμερ τώρα για τη μείωση της στόχιας. Αυτή δεν είναι, αυτή δεν είναι η ναι, ναι, έκθεση. Ναι, και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο η πορεία προς τα εμπρός. Κυρία Τσίμερ, έχετε το λόγο. Ähm, um, um Πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης, που έχει σαν τίτλο «Έκθεση για τη μείωση της ένδυας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε αναπτυσσόμενες χώρες, ο δρόμος προς τα εμπρός, τα πρόσω». Επειδή εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης, είχα την ευκαιρία να δω ποια ήταν και η αντιμετώπιση αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης και το κλίμα που επικρατούσε. Την παρουσίασα χθε και διεπίστωσα ότι εμείς ως Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόλησης θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μία γνωμοδότηση για μία έκθεση στην οποία εγώ πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό, βάσει της δικής μας εμπειρίας, βάσει αυτών που γνωρίζουμε ως πολιτική απασχόλησης, και είμαστε εμπειρογνώμονες για τα θέματα της ακαταπόλεμησης της ένδυας και της κοινωνικής πολιτικής, θα ήταν χρήσιμο να υποβάλουμε μια σειρά από προτάσεις. Το σημείο εκκίνησης, το οποίο θα ήθελα να σας υποβάλω, είναι και πάλι η συζήτηση για την έννοια της ένδυας αυτή καθεαυτή. Γιατί κατά την άποψή μου είναι κατεπηγόντως απαραίτητο ιδίω έναντι των αναπτυσσομένων χωρών και της κοινωνικής του ανάπτυξης, να τονίσουμε ότι η ένδια είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Δεν είναι μονάχα η πείνα, η έλλειψη στέγασης, η έκθεση στις ασθένειες και μόνο, αλλά ότι η ένδια θα πρέπει να ερμηνευτεί με ένα ευρύτερο τρόπο ως η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα αποδεκτό βιωτικό επίπεδο. Θέλουμε εμείς να υπενθυμίσουμε ότι στην κοινωνική διάσκεψη, την παγκόσμια διάσκεψη για τα κοινωνικά θέματα το 1995 είχαμε θεσπίσει συγκεκριμένε προτάσεις και κριτήρια. Το προηγούμενο Φεβρουάριο όταν παρουσιάστηκε η έκθεση του ΟΗΕ για την κοινωνική κατάσταση στον κόσμο υπήρξε και μια συζήτηση και πάλι για την έννοια της ε, ένδυας και έγινε σαφές ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε καλύτερα την έννοια της ένδυσης, να έχουμε μια επανεξέταση της στρατηγικής μας με σαφέστερα κριτήρια και να τη συμπεριλάβουμε στη γενικότερη συζήτηση σε σχέση με την ανάπτυξη και αυτό επομένω μα αφορά εμά και ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη και ενδιαφέρον για αυτά που γίνονται στι αναπτυσσόμενε χώρε και γι' αυτό θα πρέπει και εμεί να συμβάλλουμε στο να υπάρξει μια καλύτερη διατύπωση αυτή τη έννοια. Αυτό με οδήγησε να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σημείο και σε σημεία όπως παραδείγματος χάρη η Παγκόσμια Συμφωνία για την Δημιουργία Απασχόλησης που προτάθηκε ήδη από εμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που είχε σαν στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στις ε, συνθήκες εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όπου εμείς ε, τονίζουμε ότι πρέπει αυτή η στρατηγική να εξυπηρετήσει και την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας του ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν είναι για τη, η γνωμοδότηση που εγώ προσπάθησα να συνοψίσω εδώ. Προφανώς έχουμε περιορισμένο αριθμό σελίδων και παραγράφων που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά θα ήθελα μέσα σε αυτή τη γνωμοδότηση να θέσω τα σημεία που σας ανέφερα στο κέντρο της προσοχής μας και εγώ θα ήθελα από τη δική μου πλευρά να σας πω ότι έχω αν θέλετε ένα, μια σχεδόν ανεξάρτητη δεξαμενή από προτάσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και αν το θεωρήσουν χρήσιμο οι συνάδελφοι μπορούν με τις δικές τους προτάσεις να προκαλέσουν μια συζήτηση και εγώ φυσικά από αυτά τα οποία θα αναφέρουν θα επιλέξω ποιες από τις πολλαπλές αυτές προτάσεις θα μπορούσαμε να τονίσουμε προς την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης, γιατί ένα παρεπεραιτέρω θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα του κοινωνικού συστήματος ασφάλειας, ασφάλισης, το οποίο πρέπει να παίξει ένα ισχυρότερο ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες για την καταπολέμηση της ένδυας και ενδεχομένως θα ήταν ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά. 80% των ανθρώπων στον κόσμο, στον πλανήτη μας, δεν καλύπτονται από ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό κάνει ιδιαίτερα οξύ και πρόδειλο αυτό το πρόβλημα. Ε, επίσης θα ήθελα να επιστήσω τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Νομίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι 17 Απριλίου, εάν δεν απατώμε και θα καλωσόριζα και την συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες για τη βελτίωση αυτής της ε, γνωμοδότησης για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες ώστε να είναι μια κοινή θέση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και να γίνει σαφής η στάση μας εναντί αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. <clears throat> Στάινμπροκ, η κυρία Ζήπελ, η οποία δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα, μου ζήτησε εξ ονόματος της να δώσω την άποψή της για τα θέματα αυτά. Η κυρία Ζίπελ θεωρεί ότι είναι πολύ καλή η πρόταση της κυρίας Τσίμερ και συμφωνεί με το περιεχόμενό της, αλλά θεωρεί ότι ελείπουν ορισμένα στοιχεία από το πρώτο σχέδιο αυτής της γνωμοδότησης που θα προσπαθήσει να εισαγάγει με μία σειρά από τροπολογίες το θέμα της νομικής και οικονομικής κατάστασης των γυναικών στις χώρες αυτές, θέματα όπως η παιδική εργασία, η κατάσταση των συνδικάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όλα αυτά για την κυρία Ζίπελ είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο να είναι παρόντα στη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόκκινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Σήμερα ε, χαίρομαι που είμαι εδώ, δεν το έχω συζητήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα θα ε, πρέπει να πω ότι καταρχήν συμφωνώ με τις βασικές αρχές που θέτεται για το θέμα της μείωσης της φτώχειας και με όλες τις προτάσεις που έχετε ειδικά στο σημείο 3 όταν ε, μιλάτε για την εκπόνηση ενός χρονοδιαγράμματος καταλαβαίνω επίσης τι εννοείται για ορισμένους προδιο... Ε, περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν και τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ίσως σε ορισμένες από αυτές τις απόψεις που παρουσιάζει χρειάζεται να μπορούμε να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα και η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει προτείνει διάφορα πράγματα όπως το θέμα των μικροπιστώσεων συγκεκριμένα. Ε, είναι ένα σημαντικό θέμα για να ενθαρρυνθούν οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση των μικροπιστώσεων και συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια που ότι πρέπει κάτι να γίνει, ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε για την παιδική εργασία και μπορούμε ίσως να το εντάξουμε εδώ. σε γενικές γραμμές ε, είμαι υπέρ των όσων προτείνεται εδώ. Κυρία Μοράλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση είναι πληρέστατη, είναι εξαιρετική. Υπάρχει ένα σημείο πάνω στο οποίο ε, πραγματικά δεν ε, βρήκα αυτά που περίμενα Πρόκειται για τις γυναίκες, για τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση παινίας εξαιρετικά μεγάλη γιατί μόλις χειρέψουν χάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους και ε, εφόσον θέλουμε, έχουμε σαν στόχο τη μείωση της φτώχειας, βλέπουμε ότι εδώ οι γυναίκες είναι οι πιο φτωχές μες τους φτωχούς και ε, εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα στη ζωή τους αυτό δημιουργεί περαιτέρω παινία στο, στην κατάσταση των γυναικών και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ειδικό θέμα. Η κυρία Ζήμερ ε, θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, υποδείξεις των συναδέλφων. Εγώ είμαι έτοιμοι να δεχτώ τις συγκεκριμένες προτάσεις τροπολογιών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και τη, τους μεμονωμένους βουλευτές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με οποιαδήποτε τροπολογία εφόσον παραμένουν συνεκτικές με το θέμα το οποίο μας ε, απασχολεί. Απλώς εγώ σε αυτή την πρώτη παρουσίαση άφησα απ' έξω το θέμα αυτό και σας δίνω απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, το θέμα ορισμένων ομάδων στόχου όπως αναφέρθηκε επαγγελματικά το θέμα των γυναικών, το θέμα της παιδικής εργασίας, το θέμα των ηλικιωμένων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ οξέα τα προβλήματα αυτών και θα πρέπει εδώ να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτούς. Υπάρχει λοιπόν μια, ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων και θα πρέπει με τη συζήτηση με τα μέλη αυτής της Επιτροπής να μπορέσουμε να δούμε ποια ακριβώς θα είναι τα στοιχεία αυτού του φάσματος τα οποία θα προβάλλουμε στη χνομοδότησή μας. Ε, θα υποβάλω και τροπολογίες για τους ανθρώπους με δικές ανάγκες. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 7η Απριλίου, μεσημέρι, 28 Απριλίου η οθέτηση, ε, στις 10 Μαΐου θα ευθυθεί στην ΤΕΒΕ και μάλλον στην Ολομέλεια του Ιουλίου θα υιοθετηθεί το θέμα.